Thank you very much. I open the meeting of Committee. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Περιφερειών σήμερα το απόγευμα και αύριο όλη την ημέρα. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Έχετε μήπως σχόλια? Είχαμε κάποιες αλλαγές ε, τελευταία στιγμή σε αυτή την ημερήσια διάταξη, αλλά νομίζω ότι δέχτηκαν όλοι τις αλλαγές αυτές. Μάλιστα, πολύ ωραία. Επόμενο σημείο, η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 3ης Σεπτεμβρίου και της 13ης Σεπτεμβρίου. Έχουμε τα σχέδια των πρακτικών της 3ης και της 13ης Σεπτεμβρίου online ως ήθιστε. Προτείνω ε, εκτός αν, δεν, έχετε αντιρρήσεις που θα εκφράσετε στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, να θεωρήσουμε πως εγκρίνονται. Δεν υπάρχουν σχόλια. Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχω μόνο μία ανακοίνωση, ότι δηλαδή πρέπει να σας ενημερώσω ότι έγινε μία ε, συνεδρίαση ανάμεσα στην Επιτροπή ε, στη διάσκεψη των Προέδρων και το επιτρόπους, ε, την ομάδα των επιτρόπων, έγινε στη Στρασβούργο. Ήθιστε κάθε Οκτώβριο να γίνεται μια συνεδρίαση, μάλλον κάποιες συνεδριάσεις, ώστε να συζητηθεί το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για την επόμενη χρονιά. Φέτος η συνεδρίαση αυτή έγινε στις 2 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο πέντε συνεδριάσεις με διάφορες, διάφορους σχηματισμούς προέδρων των Επιτροπών και Επιτρόπων ανάλογα με τα θέματα, τα χαρτοφυλάκια ε, μαζί με τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης. Εγώ συμπροείδρευσα στην συνεδρίαση που είχε αφιερωθεί στην συνοχή και τις αξίες όπου συζητήσαμε έξι επίτροποι και δέκα πρόεδροι των επιτροπών ε, και συζητήσαμε για πολλά και διάφορα θέματα. Θα πρέπει να πω ότι ήταν ο κύριος Ντομπρόφσκης, ο κύριος Κατάινεν, είχαμε τον επίτροπο για ε, την παιδεία, για τις κοινωνικές υποθέσεις, τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για το κράτος δικαίου και η συζήτηση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η σειρά των συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε με μια ολομέλεια το απόγευμα, στην οποία συμπροείδευσαν ο κύριο ε, Τίμερμαν και η κυρία Βίξτρομ. Κάθε ένα από του συμπροέδρου των διαφόρων ε, ε, συνεδριάσεων ανέφερε τα όσα έγιναν εκεί. Στη δική μου αναφορά τόνισα δύο βασικά πολιτικά θέματα το χρονοδιάγραμμα που πιέζει τώρα για το Ευρωκοινοβούλιο λόγω της αργοπορημένης παράδοσης της πρότασης ε, από την Κομισιόν και οι προσπάθειές μας να είμαστε όσο γίνεται πιο γρήγοροι αλλά και αποτελεσματικοί ταυτόχρονα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε την ποιότητα της ε, της εργασίας μας και της απόφασής μας στη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά Επίσης ανέφερα πως η διαδικασία και η χρονική πίεση θα συνεχιστούν και μετά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία μετά τις εκλογές και οφείλουν να είναι τόσο δραστήριοι και επιμελείς μέχρι την τελευταία μέρα της εντολής τους όσο και εμείς γιατί και εμείς προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο δραστήριοι, πιο ενεργοί και να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο για να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Η Κομισιόν θα πρέπει να πράξει το αυτόν μέχρι την, το πέρας της εντολής της. Το δεύτερο θέμα που τόνισα ήταν η συζήτησή μας για το πρόταση περί κράτους δικαίου. Το θέμα που ήθελα εγώ να καταστήσω σαφές ήταν ότι το κράτος δικαίου δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεχωριστεί από τα ευρωπαϊκά μέσα και προγράμματα που προωθούν τις επενδύσεις την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Αντιθέτως αποτελεί ένα απαραίτητο πλαίσιο εντός του οποίου εργαζόμαστε και μέσω του οποίου δημιουργείται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η συσχέτιση ανάμεσα στο κράτος δικαίου και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και την προστιθέμενη αξία θα πρέπει να είναι σαφής και, κατανοώ, και κατανοητή από τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα για τις ευρωεκλογέ. Αυτά λοιπόν συζητήσαμε. Επίτροπος Κρέτσου ήταν επίσης παρούσα και ενημέρωσε τους επιτρόπους ε, και τους πρόεδρους των επιτροπών για τις προτάσεις τους. Εμείς έπρεπε να ενημερώσουμε τους πάντες για το χρονοδιαγραμμά μας και για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Ποια, είναι η αλήθεια ακριβώς, γιατί ακριβώς κινούμαστε με πολύ καλό ρυθμό στα βασικά μας θέματα. Αυτά λοιπόν έγιναν σε εκείνη τη συνεδρίαση. Δεν συζητήσαμε το μελλοντικό ε, πρόγραμμα, διότι δεν έχουμε δει πρόγραμμα για το 2019. Έχουμε ε, δει ποιες είναι οι ευθύνες της Επιτροπής στη συνέχεια ε, στην ακολουθία της εργασίας της και πλήρη υποστήριξη προς το Κοινοβούλιο υπάρχει για πιο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτά λοιπόν ήταν οι ανακοινώσει μου. Και τώρα περνάμε στο τέταρτο και κύριο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης. Αποφάσισα να φιερώσουμε ολόκληρη μας τη συνεδρίαση σχεδόν απόψε σε λεπτομερή εξέταση του σχεδίου έκθεσης της πρότασης της Επιτροπής για το κοινό κανονισμό για την περίοδο 2021 μέχρι και 2027. Πρόκειται για ένα, μια πρόταση νομοθετική που σχετίζεται με το PDP και είναι πολύ μεγάλης πολιτικής σημασίας για την Επιτροπή μας καθώς θεσπίζει του τους κύριους κανόνες για τη μελλοντική περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχή. Η πρώτη παρουσίαση και συζήτηση με την Επιτροπή έγινε στις 20 Ιουνίου. Εδώ οι εισηγητέ έκαναν διάφορες προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για βασικά θέματα με την Επιτροπή και η Γραμματεία και την γραμματεία που στηρίζει τους συνεισηγητές, όπου ε, μάλιστα έγιναν διάφορες τεχνικές ε, συνεδριάσεις, ε, τεχνικές γνώσεις, παρουσιάσεις powerpoints, πρακτικά των συζητήσεων, μελέτες και ενημερώσεις που προετοιμάστηκαν από τις ερευνητικές υπηρεσίες έχουν δοθεί σε όλους τους κοιόδες εισηγητές μας και στους πολιτικούς συμβούλους μας. Σήμερα οι συνεισηγητές, η κυρία Κρέλ και ο κύριος Νόβακοφ, ε, υποβάλλουν το σχέδιο έκθεσής τους. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους εισηγητές, στη συνέχεια στους κοιόδης και μετά στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών. <clears throat> Μετά θα ακούσουμε και την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, των Περιφερειών που θα μας την υποβάλει η κυρία Μαρίνη που θα είναι εδώ παρούσα και θα μας το παρουσιάσει εδώ στην ε, αίθουσά μας. Αλλά μαζί μας σήμερα είναι και ο κύριος Μπος Ρόιτ που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή και Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και είναι εισηγητής για τη δική τους νομοδότηση για το ίδιο θέμα και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και την θέση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Αυτό λοιπόν, έτσι θα έχει λοιπόν η συνεδρίασή μας και δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Κρέλ. Σας ευχαριστώ θερμά κυρία Πρόεδρε. Πράγματι ήταν δύσκολες οι εβδομάδες και οι μήνες εκείνοι κατά τους οποίους ε, προετοιμάσαμε αυτήν την κοινή έκθεση έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό και προκειμένου να επιτύχουμε τον ενδιάμεσο στόχο της ε, ψήφισης αυτής της έκθεσης ε, τον Δεκέμβριο αυτού του έτους έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει και η ψηφοφορία τον Ιανουάριο ε, και προκειμένου έτσι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Ε, νομίζω πως ε, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι περιφέρειες να εμπλακούν όσο το νωρίτερο δυνατό στην όλη διαδικασία του σχεδιασμού και, στη, και της διαχείρισης. Και έτσι λοιπόν σε αυτό θα συμβάλλει ακριβώς το να έχουμε καταρχήν ένα αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις δικές μας διαπραγματεύσεις. Ε, και ελπίζουμε πω ε, και η Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων θα επιδείξουν και εκείνη μια επικοδομητική στάση. Ε, εγώ θα κάνω μια αρχή εδώ στην παρουσίασή μου και ο συνάδελφος Νόβακοφ θα συνεχίσει με την παρουσίαση των βασικών αλλαγών που προτείνουμε εμείς σε αυτή την πρόταση της Επιτροπής με την έκθεσή μας. σε ό,τι αφορά το σύνολο της διαρθρωτικής ε, πολιτικής, η πιο βασική αλλαγή την οποία προτείνουμε σε σχέση πάντοτε με την πρόταση της Επιτροπής είναι ότι σε όλα τα άρθρα όπου αυτό είναι απαραίτητο ουσιαστικά συμπεριλαμβάνουμε και πάλι υπό την αιγίδα, αν θέλετε, του γενικού κανονισμού τα γενικά κονδύλια από το Γεωργικό Ταμείο στο Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξη. Ε, ε, αυτό το γνωρίζετε και από πριν ότι σκοπεύαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και οι σχετικέ συζητήσει ήταν πολύ θετικέ. Ε, και Ε, βέβαια, η Επιτροπή είχε καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα, δηλαδή στο να βγάλει από τον γενικό κανονισμό η Επιτροπή αυτό το Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξη. κάτι. δική μα άποψη, δεν είναι σωστή αυτή η απόφασή τη. Αντιλαμβανόμαστε αυτό σκεπτικό ότι δηλαδή θέλουν να, να, να έχουν αυτά τα ταμεία του πρώτου δηλαδή και του δεύτερου ε, πυλώνα στο, ε, υπό την ίδια αντιμετώπιση, αλλά εάν θέλουμε ε, εμείς από τη δική μας πλευρά να συμπεριλάβουμε και πάλι το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο γενικό κανονισμό δεν σημαίνει ότι θα ε, ουσιαστικά παραπέμπουμε τις σχετικές αρμοδιότητες σε όλους τους περιφερειακούς ε, υπουργού. Όχι, παραμένουν υπεύθυνα τα Υπουργεία Γεωργίας με τη μόνη διαφορά ότι στο γενικό κανονισμό υπό τον οποίο δηλαδή υπάρχουν τα ταμεία ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που σημαίνει ότι μπορούν να συνδυαστούν με πολύ καλύτερο τρόπο ε, μεταξύ τους αυτά τα ταμεία είναι πιο συνεκτικά και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την υποστήριξη όχι μόνο των ε, γεωργών σε ό,τι αφορά ακριβώ την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη τη υπαίθρου, αλλά το σύνολο ουσιαστικά αυτού ακριβώ του ε, ε, υπαίθριου χώρου, αυτών των υπαίθριων χώρων. Και θεωρούμε πω η δική μα λοιπόν πρόταση είναι πολύ σωστή και ελπίζουμε πώ θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη από εδώ από την Επιτροπή μα. Και βέβαια σε τελική ανάλυση και από την Επιτροπή Γεωργίας έτσι ώστε να δούμε ε, και να διασφαλίσουμε την εντολή της Ολομέλειας τον Ιανουάριο. Ε, στις δικές μας τώρα στροπολογίες έχουμε λάβει υπόψη μας μία πρώτη ε, εκδοχή της πρότασης που είχε προετοιμάσει η Επιτροπή για την πρόταση αυτή δηλαδή κανονισμού και η οποία μας βοήθησε και η οποία λάμβανε υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Άρα λοιπόν μία σειρά από τροπολογίες βασίζονται σε εκείνη την πρώτη εκδοχή και γι' αυτό ε, βέβαια με βάση τις αλλαγές που κάναμε και προτείνουμε στα άρθρα υπάρχουν και μία σειρά από αλλαγές της αιτιολογικής ε, σκέψης οι οποίες προκύπτουν. Μετά ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω και εδώ ακολουθώ λίγο και τη σειρά των άρθρων είναι η τροπολογία στο άρθρο 10 ότι δεν θέλουμε να έχουμε κάποια μεταβίβαση ε, προς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Invest EU. Θα θυμόσαστε ε, κατά την τελευταία ε, συνεδρίαση μας και στην σχετική γνωμοδότηση που είχαμε προετοιμάσει ακριβώς για το Invest EU είχε γίνει μια πολύ έντονη συζήτηση και να σας εξηγήσω λοιπόν το γιατί προτείνουμε εδώ αυτήν την τροπολογία για το άρθρο 10. Γνωρίζετε πως η πολιτική συνοχή στην πρόταση της Επιτροπής ε, πρικοδοτείται με 10% λιγότερα κονδύλια στο πλαίσιο του προπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη ε, θα υποστούν ε, πολύ σημαντικές περικοπές στα σχετικά κονδύλια τους. Η Επιτροπή προσπάθησε βέβαια να περιορίσει αυτές τις μειώσεις, αυτές τις περικοπές αλλά η πρότασή της έτσι όπως έχει υποβληθεί αυτή τη στιγμή με τους εθνικούς φακέλους, αυτά τα national envelopes και τις σχετικές εκλίδες κατανομής, είναι αριθμοί με, οι οποίοι ουσιαστικά οδηγούν τα κράτη-μέλη στο να πρέπει να είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίσουν στο μέλλον ε, περικοπές ε, της τάξης του 25%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να σχεδιάσουμε μια σύγχρονη πολιτική συνοχή, η οποία δηλαδή πραγματικά θα συμβαδίζει με τους σημερινούς καιρούς αλλά ταυτόχρονα μια πολιτική η οποία θα διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια. Άρα λοιπόν εμεί προσπαθούμε εδώ να διασφαλίσουμε και πάλι τα κονδύλια που είχαν αρχικά προβλεφτεί για αυτό το τομέα. Αυτό που εμεί δεν ε, στο οποίο δεν αφαρόμαστε στις δικές μας προτάσεις είναι η συνεργασία μεταξύ του InvestEU ε, και της ε, ε, και τα ταμεία του κανονισμού, γιατί στο πλαίσιο του κανονισμού Omnibus είχαμε κάνει μια σχετική συζήτηση πέρυσι και υπήρξε μια ευρεία υποστήριξη από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είναι σημαντικό αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία ε, να είναι δυνατόν να συνδυάζονται, να συνεργάζονται εύκολα μεταξύ τους. Ε, και σε συνεργασία με το Συμβούλιο μάθαμε ακριβώς ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία διαπαφής, αν θέλετε, μεταξύ των ταμείων. Και διαπιστώσαμε, για παράδειγμα, ότι σε ό,τι αφορά αυτή τη συνεργασία μεταξύ ΕΦΡ και ε, το επενδυτικό σχέδιο του ε, Πρόεδρου Γιούνκερ ήταν δυνατόν να διασφαλίζεται χρηματοδότηση διαφόρων project της τάξης έως και 100%. Πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά δηλαδή την εξασφάλιση της εθνικής συγχρηματοδότησης. Άρα λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντικό το να διασφαλίσουμε στα ίδια επίπεδα τον υφιστάμενο προπολογισμό και γι' αυτό προτείνουμε μία μεταβίβαση της τάξης των 10 δισεκατομμύρων ευρώ. Αυτή η πρόταση δηλαδή που γίνεται από το Ταμείο Συνοχής προς το You να διαγραφεί αυτή η μεταβίβαση. Και μας ε, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στην ε, ε, πρόταση της Επιτροπής ε, υπάρχει μείωση του Ταμείου Συνεχής κατά 45% αλλά το ίδιο κονδύλι προβλέπεται για, την, ε, για το μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη, το Connecting Europe Facility, το οποίο μας, δεν μας φαίνεται λογικό και μάλιστα μας φαίνεται περιττό, γιατί και η Επιτροπή μας είχε μπει κατά τελευταία συζήτησή μας ότι στο πλαίσιο τη επόμενη περίοδου χρηματοδότησης η χρηματοδότηση δεν θα γίνεται πλέον με αυτόν τον τρόπο. Θα προέρχεται δηλαδή από διαφορετικέ πηγέ και όχι από το Ταμείο Συνοχή. Η χρηματοδότηση πάντω του, του Μηχανισμού Συνδέοντα στην Ευρώπη. Αυτέ λοιπόν είναι τρει πολύ βασικέ αλλαγέ τι οποίε προτείνουμε στι ε, τροπολογίες τροπολογίε μα. Και δεν θέλω βέβαια να αναφερθώ στα πάντα γιατί ο συνάδελφο Νοβακόφ θα ε, πει και εκείνο δύο λόγια. Πάντως ε, θεωρώ πω σε γενικέ γράμμε εκείνο το οποίο θεωρώ πολύ θετικό στην πρόταση της Επιτροπής είναι το ότι δίνεται συνέχεια και βελτιώνεται ακριβώς αυτή η διαδικασία της απλούστευσης των διατάξεων. Ωστόσο, προτείνουμε μία σειρά από περαιτέρω αλλαγές εδώ του κανονισμού έτσι ώστε ακριβώς να ενισχύσουμε αυτό το στοιχείο της απλούστευσης. Ε, και η έκθεση βέβαια του ελεκτικού ε, συνεδρίου τις προηγούμενες εβδομάδες καταδεικνύει ακριβώς ε, το ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των σφαλμάτων. Ακριβώς αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δείξουμε περισσότερη εμπιστοσύνη απέναντι στα κράτη-μέλη, απέναντι στις ε, ε, περιφέρειες έτσι ώστε να επιτύχουμε τελικά και περισσότερη απλούστευση. Βέβαια, εκείνο το οποίο θα προκαλέσει περαιτέρω, περαιτέρω συζητήσει ε, ε, είναι το άρθρο 15 και η σχέση τη ε, πολιτική συνοχή αφενό με το ευρωπαϊκό εξάμεινο αφετέρου μέσω ενός νέου είδους συστάσεων αναχώρα, country specific recommendations. Νομίζω πως σε, σχέση με αυτό το σημείο θα υπάρξουν μία σειρά από προτάσεις από τους συναδέλφους, ερεθίσματα για σκέψη και βέβαια θα εξαρτηθεί μετά από τη σοφία αν θέλετε, αλλά και από την ε, διπλωματία των συνσηγητών και των σχεδόν εισηγητών, το να φτάσουμε σε μια ε, συμφωνία. Επίσης, το ίδιο διακαέστηκε και το ζήτημα των μακροοικονομικών ερεσιμοτήτων ε, και πάλι στο άρθρο 15, στο δεύτερο τμήμα του άρθρου 15. Εδώ λοιπόν αυτές οι ερεσιμότητες ή μάλλον τα σχετικά μέτρα προτείνονται ακριβώ σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι σχετικές μακροοικονομικές αρεσιμότητε από την πλευρά των κρατών μελών. Εκεί δηλαδή προβλέπονται συγκεκριμένε κυρώσει, ορισμένε διαγραφέ, για παράδειγμα κονδυλίων, επειδή για παράδειγμα ένα κράτο μέλο έχει προβεί σε κάκο διαχείριση των σχετικών κονδυλίων. Πρόκειται για δύο διαφορετικά στοιχεία βέβαια τα οποία είναι δύσκολο να συνδυαστούν μεταξύ του. Ε, η Επιτροπή επιχειρεί να το κάνει, αλλά για μα ακριβώ τίθεται πάλι το, το ζήτημα του να τα διαχωρίσουμε περισσότερο και εδώ έχουμε βασιστεί σε μία μελέτη της ε, επιστημονική ε, υπηρεσία του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να προβλέπουμε εδώ στην πρόταση κανονισμού μόνο υποχρεώσεις και όχι διαγραφή κονδυλίων και επίσης ακριβώς ακολουθώντας το πνεύμα της ε, πολιτικής ε, συνοχής, δεν θέλουμε να τιμωρούμε, να επιβάλλουμε κυρώσεις σε περιφέρειες, ε, οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν από την πλευρά τους να επηρεάσουν σε κανένα βαθμό, σε ελάχιστο βαθμό τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Άρα λοιπόν δεν θέλαμε να υπάρχει, να προβλέπεται τέτοιου είδους διαγραφή κοντιλίων. Επίσης, ε, ομολογώ ότι σε πολλές συζητήσεις που έγιναν είχα ε, λάβει την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ πιο αναλυτικοί. Για παράδειγμα, και να είμαστε και ακόμα πιο εμφατικοί και να εξαιρέσουμε εντελώς από τέτοιου είδους ε, κυρώσεις το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Αλλά το οποίο αυτή τη στιγμή εμεί δεν θίγουμε στη δική μα ε, έκθεση. σε αντίθεση τώρα με την πρόταση της Επιτροπής, εμείς προτείνουμε να επανεισαχθούν εδώ στον κανονισμό τα μεγάλα project, τα μεγάλα έργα. Ε, αυτό προκύπτει σε συνέχεια της διαδικασίας για τον κανονισμό Omnibus ε, και τη συζήτηση που είχε γίνει σχετικά, γιατί είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να, να, είναι χρήσιμο για τα κράτη-μέλη να ε, χρησιμοποιούν τέτοιου είδου ε, ειδικέ διαδικασίε σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα, τα big projects. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε πώ ακριβώ θα διαμορφωθούν οι εν λόγω διαδικασίε, αλλά νομίζω ε, πω ε, η λύση στην οποία είχαμε φτάσει στο πλαίσιο του κανονισμού Omnibus ήταν μια καλή λύση και γι' αυτό κι εμεί ω συζητητέ περιλαμβάνουμε αυτό το στοιχείο των big projects μέσα στην δική μας ε, έκθεση. Νομίζω πως είναι απόλυτα σαφές ότι σε όλες τις ε, διαπραγματεύσεις ε, τις οποίες αναφερόμαστε εμείς εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει σημαντικό ρόλο και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά και σε ό,τι αφορά το καθορισμό των μακροοικονομικών ορισμοτήτων, αλλά και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα τονίζουμε και πάλι στις δικές μας τροπολογίες και νομίζω πως ήρθε η ώρα να δώσω το λόγο στον συγητή, στο συνάδελφο, γιατί αποφασίσαμε έτσι να μοιραστούμε λίγο τις παρεμβάσεις εδώ και όλα τα στοιχεία που εγώ δεν ανέφερα μέχρι τώρα καταναφέρει ο συνάδελφος Νοβακόφ, ο οποίος είχε και τις σχετικές ιδέες για τις αναλογοτροπολογίες. Παρακαλώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου για την ε, ευκαιρία που μου δώσατε να συνεργαστώ με την Ε, Πραγματικά ήταν ε, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και είχαμε πολύ καλή συνεργασία για αυτή τη τόσο σημαντική έκθεση. Ε, μάλιστα πρόσφατα γιορτάσαμε τα 30 χρόνια της πολιτική συνοχή. Πριν από 30 χρόνια η Ευρώπη ήταν ένα όνειρο σε πολλά από τα κράτη-μέλη τα σημερινά. Ξέρω γιατί έζησα και εγώ αυτό το όνειρο. Ε, παλιά στη χώρα μου η Ευρώπη ήταν... Ε, ε ακουγόταν μόνο στις ειδήσει, στη τηλεόραση, διαβάζαμε για αυτή στις εφημερίδες. Ε, και μάλιστα στη τηλεόραση στα μεταμεσονύχτια σοου. Ε, Σήμερα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι ένα, ε, μια αίσθηση που έχουμε. Ε, δεν είναι ειδήσει ε, και τα νέα. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί πολίτες κάθε μέρα ξυπνάνε σε σπίτια που τροφοδοτούνται με αποδοτικές μορφές ενέργειας χάρη στην Ευρώπη και πολλά άλλα που είναι επιτεύγματα της Ευρώπης πολλοί ε, ε πολλές επιχειρήσεις υποστήριχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δημιουργήθηκαν επιχειρήσεις χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πολιτική συνοχή της Ευρώπης που βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματά της. Τώρα έχουμε 100 σελίδε ε, για την μελλοντική συνέχεια αυτής της πολιτικής. Και είναι στο χέρι μας ε, εμείς που δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα, να αποφασίσουμε πώς θα ε, γράψουμε τη συνέχεια αυτού του βιβλίου, είτε ως γραφειοκράτες, είτε ως οραματιστές. Η Κωνσταντζε ήδη αναφέρθηκε σε κάποιες από τις τροπολογίες που έχουμε προτείνει και είμαι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσουν με τη δική σας υποστήριξη να έχουμε καλύτερες θέσεις κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου στη συνέχεια. Ναι, κάποιες από αυτές τις προτάσεις ε, σημαίνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Συνολικά οι προτάσει μα σημαίνουν επιπλέον 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτή η Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο πολλέ φορέ σε πολλά έγγραφα, σε ομιλίε, σε ακροασει, έχουν τονίσει ότι όποιε και αν είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε, όποιε και αν είναι οι νέε πρωτοβουλίε, δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την τις παραδοσιακές και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές πολιτικές μας. Και ε, υπήρχε το σχέδιο Juncker, τώρα το έχουμε invest EU, που θα έχει συνεισφορά από την πολιτική συνοχή. Μετά έχουμε την, ε, το Ευρώπη ορίζοντας, το συνδέοντας την Ευρώπη. Κάθε φορά είναι κάτι καινούριο. Το να είμαστε προσεκτικοί στις μεταφορές ε, που γίνονται από εδώ και εκεί δεν σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι με τις πρωτοβουλίες αυτές, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι υποστήριξή τους και όχι παίρνοντας χρήματα από την, ε, ε, από την πολιτική συνοχής. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το 85% για τις ε, λιγότερο επιτυχημένες περιοχές, 70% για τις μετάβασεις και αντίστοιχα για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Ε, αυτό είναι που θα ε, μας ε, κάνει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Τώρα για το θέμα των ε, μεταφορών από ε, ένα πρόγραμμα σε άλλο και για την χρήση της πολιτικής συνοχής για να χρηματοδοτήσουμε άλλες πρωτοβουλίες. Είναι σαν να παίρνουμε τούβλα από ένα σπίτι και να το χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε ένα άλλο σπίτι. Σαν αποτέλεσμα δεν θα είναι κανένα από τα δύο σπίτια όμορφο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λοιπόν να υποστηριχθούν αυτές οι άλλες πρωτοβουλίες, αλλά όχι από την πολιτική συνοχή. Ε, ίσως θα θυμάστε την περασμένη φορά που είπα στις αρχές του καλοκαιριού, όταν συνεργαζόμουν με την Κωνσταντσε, ότι θα πρέπει να συντάξουμε μια, ένα σχέδιο έκθεση που να είναι εύκολο να το διαβάσει κανείς, να διαβάζει μια εφημερίδα και που θα μας βοηθήσει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτή η απλούστευση είναι κάτι που δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε ε, για κανένα λόγο. Γιατί οι περισσότεροι δικαιούχοι αυτό που, που μας λένε πρώτα απ' όλα ε, και πριν απ' όλα είναι το να κάνει κανείς αίτηση για συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι όσο απλό είναι να παραγγείλεις ένα καφέ σε μια καφετέρια. Τις περισσότερες φορές, και το έχω αναφέρει αυτό πολλές φορές στις συναντήσεις μας, ε, σε υπουργού που είναι υπεύθυνοι για την περιφερειακή ανάπτυξη, σε πυρογνώμονες, ε, στις μόνιμες αντιπροσωπίες στους δικαιούχους, το ίδιο αίτημα μας απευθύνουν όλοι αυτοί. Να γίνουν τα πράγματα όσο γίνεται πιο εύκολα. Εμείς δημιουργήσαμε μία θέση που ίσως ε, απαιτεί περισσότερο χρόνο για να είναι κατανοητή σε ορισμένα σημεία. Η τεχνική βοήθεια, παραδείγματο χάρη, ναι, εγώ το θεωρώ ότι σημαίνει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν πόσο περισσότερο θέλουν και πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Άρα χρειάζεται ένας ευέλικτος μηχανισμός ε, που το κράτος μέλος θα αποφασίζει πότε και πόσο θέλει από το φάκελο τεχνικής βοήθειας κάθε φορά. Επιπλέον, το σχέδιο της Κομισιόν, και χαίρομαι που έχουμε εκπροσώπους της Κομισιόν εδώ, μιλάει για μεταφορές κονδυλίων στο Invest EU μέχρι 5% ή αιτιολογημένες περιπτώσεις μέχρι και το 100% αν το αποφασίσει το κράτος μέλος. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχω καταφέρει να καταλάβω τι σημαίνει δεόντω αιτιολογημένε περιπτώσει. Χρειαζόμαστε κάποιε εγγύησει ότι η συνοχή πολιτική για αυτό το κράτο μέλο δεν θα θυσιαστεί ακόμα και σε εθελοντική βάση. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι τελικά καταφέραμε να συμμορφούμε με το σφιχτό πρόγραμμα που είχαμε και και ελπίζω ότι θα ανταποκριθείτε από την πλευρά σας και θα δείξετε προθυμία να μας βοηθήσετε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, διατηρώντας την καλή ποιότητα της έκθεσης. Βεβαίως παραμένουμε ανοιχτοί για τα σχόλιά σας και με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Thank you. These were Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν, αυτές ήταν οι εισηγήσεις των δύο ε, εισηγητών. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδες. Η κυρία Τόμας, πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να επανέλθω σε κάποιες από τις προτάσεις των συνεισηγητών και τις υπόλοιπες μου προτάσεις θα τις υποβάλω ε, σαν τροπολογίε. Η, προ... Κομισιόν προβλέπει μία... ένα μικρότερο κονδύλι σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Εγώ στηρίζω την πρόταση των δύο συνεισηγητών ώστε να αυξηθεί κατά 12% το συνολικό ποσό, ώστε να έχουμε ένα επίπεδο αντίστοιχο με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Στην πρόταση τη Κομισιόν επίση, η προχρηματοδότηση ε, απελευθερώνεται ε, ετήσια. Όμως εγώ στηρίζω την αύξηση του ποσοστού προχρηματοδότησης μέσα στο πολιτές πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε να ε, λάβουμε υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης για όλη τη διάρκεια της περίοδου. Δεν θα πρέπει δηλαδή να τιμωρηθούν οι κοινότητες και οι τοπικές ε, ε, ενώσεις λόγω των εθνικών πολιτικών. Γι' αυτό και θεωρώ ότι όταν δεν υπάρχει αρκετή συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές συστάσεις να αναστέλλεται η καταβολή των κονδυλίων που έχουν δεσμευθεί ως υποχρεώσεις και όχι ως πληρωμές. Η επανεξέταση επίσης είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην πολιτική συνοχή διότι οι όροι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν στη διάρκεια της επταετίας. Γι' αυτό και σύμφωνα με την εμπειρία που είχαμε ε, τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι οικονομικές κρίσεις είναι από τους κύριους λόγους για τους οποίους μπορεί να αιτιολογηθεί ένας νέος προσανατολισμός των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής. Στην περίοδο 2014 με 2020 είχαμε προβλέψεις όπου εισάγονταν ε, μέτρα ειδικού ελέγχου για τα μεγάλων διαστάσεων προγράμματα. Αυτού του είδους οι διατάξεις δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν στο πλαίσιο αυτής της απόπειρας μείωσης του διοικητικού φόρτου. Ωστόσο, για τα μεγάλα προγράμματα θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και απλοποίηση των κανόνων που ισχύουν με κατόφλια ωστόσο πιο υψηλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενος σκιώδης εξ ονόματος της ομάδας ALDE είμαι εγώ και θα σας, δώσω τη γνώμη μου για το σχέδιο νομοθετικής έκθεσης για την πρόταση CPR. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο συγητές, Κρέλ και Νοβακόφ, για την προετοιμασία της έκθεσης για τον κοινό κανονισμό. Σας, σας ευχαριστώ που συνεργαστήκατε με το, με τόσο στενό ε, χρονοδιάγραμμα και υποβάλλατε μια τόσο φιλόδοση έκθεση. Θα ήθελα να υποβάλω τα εξή σχόλια για το σχέδιο ε, έκθεσης. Δεν θα καλύψω όλα τα θέματα, αλλά στα περισσότερα ζητήματα να πω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις και συμβιβαστικές. Θέλω όμως να αναφέρω κάποια από τα ε, σημαντικότερα σημεία. Το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει διάφορα κύρια σημεία, ένα εκ των οποίων είναι η επανένταξη από πλευρά των εισηγητών των σχετικών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την ανάπτυξη της Υπέθρου. Καταρχάς, στηρίζω την συμπερίληψη αυτή, όμως θέλω να τονίσω πως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον κατάλληλο συντονισμό και συνεργασία με την Επιτροπή Γεωργίας. Και επίσης να σκεφτούμε την κοινή θέση για τις δύο επιτροπές, διότι μόνο η συμπερίληψη σε τέτοιου είδους ε, κανονισμούς, χωρίς όμως σχετικά κείμενα που να περιλαμβάνονται στον κανονισμό για την γεωργία, για το Γεωργικό Ταμείο δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να έχουμε εκ των προτέρων συντονισμό. Ένα ε, κατάλληλο ε, μηχανισμό συντονισμού θα πρέπει να δημιουργηθεί από τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουμε τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ε, πολιτική συνοχή και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου στο μελλοντικό πλαίσιο. για τις περιοχές ε, τις ορεινές αλλά και τις ε, ε, περιοχές γύρω από τις πόλεις γιατί ήδη έχουμε σχετικά ψηφίσματα στην Επιτροπή Περιφερειών για περιφερειακής πολιτικής και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, είναι δική μας ευθύνη να βρούμε και να καταφέρουμε σωστό συντονισμό ανάμεσα σε όλα τα μέσα που έχουμε ε, στον τομέα αυτό. Δεύτερο κύριο στοιχείο της έκθεσης είναι η διαγραφή της σύνδεσης με το Ευρωπαϊκό Εξάμενο και τις διαρθωτικές ε, τα διαρθωτικά μέτρα και μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω αντίθετα ότι ο συντονισμός με το εξάμεινο και τις ιδιωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να τονώσουν την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών ταμείων και του κοινωνικού του Ταμείου Συνοχής. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και έχουμε διαφορετικές απόψεις. Όμως σε αυτή την περίπτωση πιστεύω πραγματικά πως όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και όταν προσπαθούμε να υπερασπιστούμε το, την πολιτική συνοχή και να βρούμε εξύγχρονη ε, πολιτική συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε κατάλληλη, ε, κατάλληλο συνδυασμό, λειτουργικό συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη χρειάζονται οι μεταρρυθμίσεις. Συσχέτιση λοιπόν με τις μεταρρυθμίσεις και τα διορθωτικά ε, μέσα, διότι έχουμε παραδείγματα όταν στηρίζουμε ένα πρόγραμμα σε κάποια κράτη-μέλη, λαμβάνεται ναι μεν η στήριξη, χωρίς όμως να έχουν γίνει απαραίτητε μεταρρυθμίσεις και ότι δεν επιτυγχάνεται εν τέλει, ε, δεν δημιουργείται μάλλον ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από αυτού του είδους τα project. Τρίτο στοιχείο είναι η διάκριση της δυνατότητας του... Του... του προγράμματος θελοντικής μεταφοράς το 5% για πολλά από αυτά τα προγράμματα από τα προγράμματα ε, στις ε, δομές της ευρωπαϊκές με άμεση ή έμεση διαχείριση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται τελείως επί θελοντικής βάσης και να εκφράζει την ευελιξία χρήσης των ε, ταμείων και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού εν γέννη. Και καλωσορίζω το κείμενο της Επιτροπής. Θεωρώ πως η ευελιξία μαζί με την απλοποίηση είναι η λέξη κλειδιά για την ε, αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της πολιτικής συνοχής. Ε, δυνατότητα λοιπόν μεταφοράς κάποιων περιορισμένων ποσών από τα δευτικά ταμεία θα στηρίξει την σωστή απορρόφηση και τα καλά προγράμματα με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ειδικά όταν μιλάμε για project διασυνοριακού τύπου. Επίσης, στηρίζω την ε, μεταφορά προς την ε, ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Γιατί αυτό, αυτή η πρόταση βασίζεται στην επιτυχή προσέγγιση του 2014 με 2020 και λαμβάνει υπόψη την σημασία των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κατασκευή των ε, κρίκων που λείπουν ώστε να λειτουργεί ε, ομαλά να λειτουργούν ομάλα τα δίκτυα. Είναι ένα από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να δημιουργήσουμε αυτά τα δίκτυα στην Ευρώπη. Εγώ εκπροσωπώ μια χώρα που είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δίκτυα και ξέρω πως υπάρχουν ε, κάποιοι στην Ευρώπη που προσβλέπουν στις καλές διασυνοριακές συνδέσεις για τις μεταφορές μιλώ. Και μια βασική λειτουργία είναι το συνδέοντα στην Ευρώπη. Θα το συζητήσουμε, είναι μια επιλογή, θα το συζητήσουμε, αλλά εγώ πιστεύω πως είναι μια που πρέπει να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο και να πάνε και κάποια, τα, κάποια χρήματα από την πολιτική συνοχή. Τέταρτο στοιχείο αφορά την αρχή της εταιρικής σχέσης και την αρχή της πολυεπίπεδης διαχείρισης, διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ που τα συμπεριλάβατε εδώ αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά για την, για την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής. Θέλω να ακούσω τη γνώμη και της Επιτροπής Περιφερειών και της ΟΚΕ ε, ε, για το κατά πόσο αυτή η αρχή της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να είναι στη βάση. Επιπλέον, θέλω να στηρίξω τις επιπλέον πόρους που προτείνονται για τη μεγαλύτερη επικοινωνία, καλύτερη επικοινωνία και ορατότητα των κονδυλίων από πλευράς του κοινού, καθώς και η συνειδητοποίηση για τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία αυτών των προγραμμάτων στήριξης. Ήδη έχουμε εμπειρία από τις διαπραγματεύσεις όμνιμπους. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί κατά τη γνώμη μας, να βελτιωθούν αυτές οι προτάσεις για την καλύτερη επικοινωνία. Γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να παρουσιάσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες την πραγματική αξία της πολιτικής συνοχής. Τέλος, ε, εφόσον πρέπει οπωσδήποτε να, αντιμετωπιστεί το, να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές σε συμφωνία με τη Συμφωνία του Παρισιού, ορίζω τον τροποποιημένο στόχο των εισηγητών για mainstreaming των περιβαλλοντικών ε, θεμάτων που θα πρέπει να φτάσουν στο 30% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της στήριξης κλιματικών στόχων. Σας ευχαριστώ και πάλι ε, προς τους εισηγητές και προσβλέπω στις ε, καρποφόρες συζητήσει μας με τους σκιώδεις εισηγητές. Αυτή ήταν η δική μου ε, παρέμβαση ως σκιώδης και τώρα προχωρούμε με τον κύριο Μαρζέ και μάλλον την κυρία Μισελ που θα παρουσιάσει την θέση της ομάδας. Ευχαριστώ θερμά κυρία Πρόεδρε και εγώ καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δύο συνεχιστητές δηλαδή την κυρία Κρέλ και τον κύριο Νόβακο γιατί θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τα βασικά ζητήματα πραγματικά οι απόψεις μας ταυτίζονται και νομίζω πως η έκθεση ε, πραγματικά ε, είναι ε, ισορροπημένη με τον σωστό τρόπο. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν έχετε την πλήρη υποστήριξη μας σε ό,τι αφορά το την επανασυμπερίληψη, αν θέλετε, του Ταμείου Αγροτική Ανάπτυξη και πάλι εδώ στον κανονισμό. Ήδη το είχαμε αναφέρει αυτό και στο παρελθόν, γιατί εμεί θεωρούμε πω ε, είναι αυτονόητο το γεγονό ότι η αγροτική ανάπτυξη αποτέλεσε πάντοτε σημαντικό στοιχείο τη ε, πολιτική συνοχή και θα, θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί στοιχείο τη. Σε ό,τι αφορά την δυνατότητα μεταβίβασης κονδυλίων ε, της πολιτικής συνοχής προς το InvestEU. Συμμεριζόμαστε την επεκριτική σας ε, στάση. Ε, είτε εδώ αναφέρεται το EFSI, είτε το InvestEU. Έχουν διαφορετικούς στόχους αυτά τα ταμεία έχουν διαφορετικά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης, άλλες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και άλλες μορφές χρηματοδότησης, οπότε τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής που ήδη ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί δεν θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω, ακόμα και αν μιλάμε για μικρά ποσοστά. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιτρέψουμε την εξαφάνιση ακόμα περισσότερων κονδυλίων από την πολιτική συνοχή. Επίση, από τη δική μα πλευρά, υποστηρίζουμε την διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία μέσω Interreg και την περαιτέρω ενίσχυσή της. Αλλά να πω πως κατά τελευταία επίσκεψη ε, της δικής μας, ε, δικής μας επιτροπής από την ε, αντιπροσωπείας από την Επιτροπή μας στην Ρεουνιόν είχαμε δει πόσο μπορούν να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα του Interreg για τέτοιου είδους περιοχές. Και φυσικά υποστηρίζετε Υποστηρίζουμε από τη δική μα πλευρά πλήρω την αξίωσή σα στα ε, κονδύλια τη πολιτική συνοχή να παραμείνουν ε, στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά. Ε, από εκεί και μετά όμω να κάνω και κάποιε συμπληρωματικέ παρατηρήσει πέρα δηλαδή από όλου του επένου αυτού. Ε, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά χρηματοδότηση, νομίζω πω θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ ε, αυτά τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ε, για συγκεκριμένε ε, περιοχές γιατί βέβαια αυτές ειδικότερα οι απομακρυσμένε περιοχέ έχουν κατηγοριοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο που σημαίνει ότι θα υπάρχουν περισσότερες περιοχές που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και άρα θα πρέπει να μοιραστούν μεταξύ τους τα ίδια κονδύλια. Ενώ σε ό,τι αφορά αυτές τις κατηγορίες έχει, είχε επιτραπεί μέχρι στιγμής σε ποστό σε χρηματοδότηση έως το 85% πράγμα το οποίο δεν συνεχίζεται στη νέα πρόταση και αντιπροτείνεται 60%. Ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, το 70% θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή ε, συμβαστική ε, λύση. Άλλωστε, μια τέτοια αναφορά κάνει και η έκθεση από την πλευρά τη Επιτροπής των Περιφερειών και μια τέτοια πρόταση και θα ακούσουμε και την παρουσίαση τη επιτροπή Περιφερειών. Ή εναλλακτικά θα μπορούσαμε ε, στο πλαίσιο μιας συμβαστική λύσης να προβλέψουμε ειδικέ διατάξει για, να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ ασφαλείας, κάτι δηλαδή που υπήρχε, υπήρχε και μέχρι στιγμή. Από εκεί και μετά, εκείνο που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε είναι ότι πολέμηση της ένδυας και των διακρίσεων όπως για παράδειγμα η δημιουργία των ε, σωστών θέσεων εργασίας ε, δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα γιατί πραγματικά συνεχίζει να είναι προτεραιότητα και αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για, τα οποία, για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί και κατά συνέπεια λοιπόν αυτοί οι στόχοι της καταπολέμησης ένδυας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ε, στους βασικούς στόχους και να αναδεικνύονται ε, στα ε, κυριότερα χρηματοδοτικά μα εργαλεία. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εξαμενού και των μακροοικονομικών αιρεσιμοτήτων, ε, η δική μας θέση είναι γνωστή νομίζω. Εξακολουθούμε δηλαδή να πιστεύουμε ότι και τα δύο αυτά θα πρέπει να τεγραφούν. Αλλά αναγνωρίζουμε βέβαια το ότι οι συγητές ήδη από τώρα προσπαθούν να προτείνουν μια συμβαστική λύση. Οπότε, Κωνσταντς, θα δούμε τελικά ποιο θα είναι το, το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, σε ποιο συμβασμό θα καταλήξουν. Σε ό,τι αφορά και πάλι αυτές τις ερεσιμότητες, πάντως ε, θα πρέπει να ισχύσουν μόνο τέτοιες οι οποίες θα είναι δυνατόν να ε, συγκαθοριστούν και από τις ίδιες τις ε, περιφέρειες. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα αιτήματα ε, των περιφερειών σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των ε, ειδικών των περιοχών N3, στόχων N3 και τη διατήρηση των σχετικών κονδυλίων υποστήριξη. Και εμεί θα προτείνουμε σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση η, ο παναπρογραμματισμός να γίνει μόνο σε, ε, θελοντική βάση και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάτι τέτοιο θα κριθεί πραγματικά απαραίτητο γιατί οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει περισσότερο γραφειοκρατικό άχθος εδώ. Αλλά νομίζω πως στην ίδια κατεύθυνση κινούμαστε όλοι μας. Και επίσης και στο πλαίσιο και πάλι της αξιολόγησης ε, του τελευταίου ταξιδιού εδώ αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας θα ήθελα να ζητήσω να αξιώσουμε ε, με πιο εμφατικό τρόπο, πιο κατηγορηματικό τρόπο τη συμπερίληψη των οργανισμών περιφερειακής τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον σχεδιασμό ε, και την κατανομή των κοντιλίων των διαφόρων ε, ε, ταμείων, γιατί νομίζω πως διαφάνει στην επίσκεψή μας στη Ρεουνιόν είναι το γεγονός ότι συχνά στην προετοιμασία αυτών των προγραμμάτων κατά τον σχεδιασμό τους δεν περιλαμβάνονται οι οργανισμοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και τα συνέπεια όλος αυτός ο σχεδιασμός γίνεται άνωθεν. Και γι' αυτό η αξίωση την οποία έχουμε επαναλάβει ξανά και ξανά, δηλαδή η έγκαιρη εκ των προτέρων συμπερίληψη σε αυτές διαδικασίες σχεδιασμού αυτών των οργανισμών είναι πολύ σημαντική. Γιατί όταν κάνουμε λόγο για αποτελεσματικότητα, τότε ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι εκταμιεύσεις αυτές γίνονται ακριβώς ε, στις κατατόπους περιοχές. Άρα λοιπόν για μας είναι σημαντικό αυτή ακριβώς η διάσταση να υπογραμμιστεί ακόμα περισσότερο. Φυσικά θα υποβάλουμε και τις δικές μας τροπολογίες, ήδη έχουμε υποβάλει κάποιες και όπως ε, και οι συγητές και εγώ στη Ιώδη συγγήτρια αναμένω με ενδιαφέρον τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ. Ε, η ε, κυρία Ντεμάτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, Νοβάκοφ και κρέλε για την πρώτη εκδοχή αυτής της έκθεσης. Πριν να περάσω σε κάποιες επισημάνσεις, θα ήθελα να ζητήσω συγκεκριμένη προθεσμία για την, ε, παρουσίαση, για την υποβολή των τροπολογιών, γιατί ε, φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα πολλές ε, ε πλευρές που πρέπει να εμβαθύνουμε, ερεσιμότητα, δείκτες κλπ. Ε, και σχεδόν πάντα η ταχύτητα είναι εις βάρος της ποιότητας. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω κάποια σημεία για μένα σημαντικά. Συμφωνώ να αυξήσουμε όσο το περισσότερο ε, τη συνέργεια ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα διαρθρωτικά ταμεία. Ε, γιατί διαφορετικά υπάρχει κινδύνος να ε, διαστρεβλωθούν οι στόχοι και η συνεισφορά αυτού του ταμείου. Συμφωνώ επίση με το σκεπτικισμό όσον αφορά τη μεταφορά κονδυλίων από τα ταμεία συνοχής στο Invest EU. Κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό να εισαχθεί έστω και αν, όπως λέει η Κομισιόν, η μεταφορά αυτή είναι προαιρετική, να υπάρχει ένας περιορισμός εδαφικός, ε, να γίνονται οι μεταφορές στην, περιφέρεια του, στην ίδια περιφέρεια του κράτους μέλους. Ε, επίσης, ε, η έννοια της εταιρικής σχέσης δεν γίνεται πάντοτε σεβαστή και θα πρέπει να ενισχυθεί. Και εδώ ε, συμφωνώ με κάποιες σχετικές τροπολογίες. Εκφράζουμε επίσης την ανησυχία μας για την ισχυρότερη, την ισχυρότερη σύνδεση που γίνεται ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ε, θυμόμαστε το άρθρο 23 του παλιού κανονισμού που είναι τώρα το άρθρο 11 ε, όπου τίθεται τέτοιοι μακροοικονομικοί όροι ε, ε, σύμφωνα με την οποία μέθοδο αναστέλλονται πρώτα απ' όλα οι αναλήψεις υποχρεώσεων αλλά και οι πληρωμές σε περιφέρειες ενός κράτους μέρους που δεν ε, σέβεται τις επιταγές της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ε, ο περιορισμό αυτό να ισχύει μόνο λοιπόν ζητάμε για τι αναλήψεις υποχρεώσεων και από την άλλη πλευρά υπάρχει υποχρέωση εκ μέρου τη Κομισιόν. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση να ενημερώνει η Κομισιόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ανασταλούν ε, οι πιστώσει αυτέ. Ε, θα υποβάλω και σχετικέ τροπολογίε για τα θέματα αυτά. Μετά, η συζήτηση για τη συγχρηματοδότηση θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη συζήτηση, λαμβάνοντα υπόψη τη σημερινή αρχιτεκτονική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης. Ε, τα η... μείωση των ποσοστών χρηματοδότηση, ας πούμε από το 85% στο 70% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, υπάρχει κίνδυνος να είναι εις βάρος των δυνατοτήτων επένδυσης. Και το ξέρουμε όλοι γιατί. Ε, υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί λόγω του Συμφώνου ε, Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, που ε, υπολογίζουν ε, τις δαπάνες, τις διαρθρωτικές δαπάνες μέσα στο ε, έλλειμμα των κρατών μελών. Από τη μια μεριά λοιπόν ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη να κάνουν μια προσπάθεια ανάπτυξης και από την άλλη ζητά από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να περιοριστούν σε αυτά τα μικρότερα ποσοστά. Τέλος, για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Αυτό αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα για την στα πλαίσια αυτής της πρότασης και τι ε, σχετίζεται πάνω απ' όλα με τον παράγοντα κίνδυνο. Δεν μπορούν να υπάρχουν κερδοσκοπικές κινήσεις και όταν υπάρχουν equity, trust fund κλπ, ε, μέσα δηλαδή υψηλής επικινδυνότητας, καταλαβαίνετε τι μεγάλο ε, κίνδυνο δημιουργεί αυτό. Πιστεύουμε ότι θα ήταν οπωσδήποτε χρήσιμο να βρεθούν τρόποι εγγύησης, αντεγγύησης ή ε, κάποια επιτόκια διευκολυντικά σε ε, εύλογα χρονικά διαστήματα ή να διευκολυνθεί το, το cloud funding, το peer-to-peer -peer to peer η και άλλοι ε, καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Καλή εργασία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν λοιπόν οι απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Ρέτσι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα για να έπαινασω κι εγώ την εργασία των δύο εισηγητών. Η εργασία αυτή ε, ε, και η έκθεση αυτή έρχονται αυτή τη στιγμή ε, στο πιο κρίσιμο σημείο κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Θα πρέπει λοιπόν να υποδεχτούμε τις θέσεις της Κομισιόν, αλλά ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε από πού ξεκινάμε. Γιατί πριν από ένα χρόνο ήμασταν εδώ και δεν ήμασταν καν σίγουροι ότι θα έχουμε μια πολιτική συνοχή προς όφελος όλων των περιφερειών. Ξέρω ότι Πολλοί λόγος γίνεται ακόμα σήμερα ε, συγκρίνονται μάλλον οι σημερινές προτάσεις που έχουμε με την τρέχουσα περίοδο. Γίνεται σύγκριση και αριθμητική μάλιστα. Δεν είναι κακό αυτό, είναι θεμητό. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν παράλληλα ένα μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην Ευρώπη εδώ και 7 χρόνια. Είναι φυσιολογικό και απαραίτητο το ξέρω, να ε, εξελιχθούν τα πράγματα, να τροποποιηθεί η πολιτική συνοχή ώστε να προσαρμοστεί ε, στα σημερινά διακυβεύματα, όπως έχουν εξελιχθεί. Και επίσης, η πολιτική συνοχή ε, έδειξε ότι ε, έχουν μεσολαβήσει ω αυτές οι εξελίξει. Κάποιε περιφέρειες που όλοι γνωρίζουμε παρουσίασαν πολύ σημαντική οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα άλλε αντιμετώπισαν σημαντικότατε δυσκολίε, επλήγησαν από βαθιά κρίση διαρκείας και επίσης ε, κάποια στιγμή κάποιες περιφέρειες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή απέναντι στις κρίσεις αυτές αναφέρομαι στο Brexit, σε άλλες προκλήσεις που εμφανίστηκαν ε, αυτή την περίοδο. Για μένα λοιπόν ε, ε υπάρχουν εδώ σημαντικά διδάγματα, όπως είπα και οι συνάδελφοι, που αφορούν την κατάσταση των περιφερειών που χαρακτηρίζονται ως σε φάση ε, μετάβασης. Ε, οι μελέτες και οι αναλύσεις μας έδειξαν ότι Κάποιες από αυτές τις περιφέρειες παρουσιάζουν και καθυστέρηση σε σχέση με τις πιο προηγμένες, πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ενώ παράλληλα τις φτάνουν οι πιο αδύναμες ε, περιφέρειες τα τελευταία χρόνια. Και έτσι οι περιφέρειες αυτές κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται απέναντι σε δυσκολίες που ε, κινδυνεύουν να αυξηθούν. Και γι' αυτό εξάλλου και η Κομισιόν πρότεινε να διευρυνθεί κατά κάποιο τρόπο η κατηγορία αυτή ε, που χαρακτηρίζεται ως ε, ε, σε φάση μετάβασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και απαραίτητο θα έλεγα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι να φροντίσουμε ούτως ώστε αυτές οι περιφέρειες οι λεγόμενες ε, να ε, επιτύχουν να επιτύχουμε να έχουν την σωστή και κατάλληλη ε, στήριξη που θα είναι στο ύψος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες αυτές για να ε, αντιμετωπίσουν αυτό τον κίνδυνο να μείνουν πίσω όπως είπαμε πριν. Και εδώ έρχεται και το θέμα του ποσοστού χρηματοδότησης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι δύο συνεισηγητές προτείνουν για αυτή την κατηγορία περιφερειών μία αύξηση μικρότερη από ό,τι για τις άλλες κατηγορίες. Γιατί η εξέλιξη είναι ε, από 70 ε, σε 65, από 55 Συγγνώμη, από 40 σε 60 για τις πιο ε, ανεπτυγμένες περιφέρειες και μόνο ε, από 50 σε 60 για τις ε, περιφέρειες μετάβασης. Εγώ συμφωνώ με αυτό που προτείνει η Επιτροπή των Περιφερειών να περάσουμε από το 60% στο 70% για αυτές τις ε, περιφέρειες σε φάση μετάβασης. Αυτό, αυτά είχα να πω. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι να συμβάλλουμε ώστε να βρεθεί μια συμβαστική λύση και μια συμφωνία που θα μας οδηγήσει σε μια ε, πολιτική συνοχή ταυτόχρονα πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο στοχευμένη. Ευχαριστώ. very much, Mr. Van Miltenburg. voorzitter. Ik zal, eh, in mijn eigen Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη δική μου γλώσσα. έτσι ώστε παρότι βέβαια θέλω να είμαι ευγενικό, προκειμένου παρόλα αυτά λοιπόν να εκφράσω την βαθιά μου απογοήτευση, γιατί νομίζω πως με αυτήν την πολιτική που εφαρμόζεται τώρα, ουσιαστικά γυρνάμε πίσω δεκαετίες. Σαν να μην υπήρχε δηλαδή καμία ε, σαν ε, να μην, υπάρχει ανάγκη για μακροοικονομικές αιρεσιμότητες, σαν να μην υπάρχει ευρωπαϊκό εξάμεινο, σαν να μην λαμβάνουμε δηλαδή υπόψη μας ε, ε, όλη την πρόοδο που έχουμε επιτύχει κατά τελευταία χρόνια και σε σχέση με πολλά άλλα εργαλεία. Γιατί βέβαια όλα αυτά έγιναν γιατί θέλουμε με κάθε ευρώ να επιτύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι θέλουμε να μείνουμε στάσιμοι και όχι απλώς να μείνουμε στάσιμοι, αλλά να υπαναχωρήσουμε κιόλας. Ε, δηλαδή, αυτά τα μεγάλα project. Γιατί κύριε Νόβακοφ δεν υπάρχει ανάγκη για παράδειγμα χρηματοδότηση στη δική σας χώρα σε χρηματοδότηση τέτοιου είδους μεγάλων έργων από αυτόν τον προπολογισμό. Και τελικά τι νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει. Δεν θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια πραγματικά συνεκτική πολιτική ε, μέσω ακριβώς των κονδυλίων που έχουμε στη διάθεσή μας, μέσω της υποστήριξης της υποδομής. Ε, δηλαδή, ακούγοντας αυτά ε, που ακούμε σήμερα εδώ, έχουμε την αίσθηση ότι η πολιτική συνοχή είναι κάτι το αποκομμένο, αλλά δεν είναι μόνη τη η πολιτική συνοχή. Υπάρχει ακριβώ για να ε, ενισχύει τι οικονομικέ και κοινωνικέ δομέ. Και ακριβώ συνοχή είναι αυτό που λείπει από αυτή την έκθεση. Ουσιαστικά προσπαθεί να ε, παραμείνει και να επιμείνει στα όσα ήδη υπήρχαν μέχρι τώρα. Και σχετικά με αυτό κάνατε και εσείς, ε, Πρόεδρε, μία πολύ καλή και σωστή παρατήρηση. Δηλαδή, εάν θέλουμε εδώ να κάνουμε αυτές τις προτάσεις, ε, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το υπόλοιπο ε, κομμάτι της ε, γεωργικής πολιτικής. Δηλαδή, σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεννοηθούμε πολύ καλά με την Επιτροπή Γεωργία. Μετά, ποσοστό προπολογισμού ε, συγχρηματοδότηση 85%. μα βρισκόμαστε ακόμα σε περίοδο κρίση, δηλαδή ειδικότερα στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία βρίσκονται ε, σε περίοδο ανάπτυξη, ε, δεν θα πρέπει να ισχύσουν χαμηλότερα ποσοστά. Αυτέ είναι οι προτεραιότητέ μα. Δεν έχουμε άλλε προτεραιότητε. Δεν υπάρχουν τα ζητήματα ασφάλεια και μετανάστευση. Θα πρέπει λοιπόν να, είμαστε, να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά επενδύουμε κάθε ευρώ από αυτά τα κονδύλια με το σωστό ε, τρόπο. Νομίζω λοιπόν πως δεν είναι ρεαλιστική η ε, προσέγγιση εδώ που ακολουθείτε. Ε, και μόνο ένα μικρό φως βλέπω στο τούνελ εδώ και θα πρέπει το αναφέρω για να κλείσω ε, θετικά τη δική μου παρέμβαση. Αυτό το 25% του ποσοστού σε ό,τι αφορά την κλιματική μεταβολή από 30% που ήταν εντάξει είναι θετικό αλλά πραγματικά είναι το, το μοναδικό σας λέω θετικό στοιχείο που βρίσκομαι πραγματικά απογοητευμένος γιατί ουσιαστικά δεν απηχεί αυτή η πρόταση, αυτή η έκθεση τα αποτελέσματα των συζητήσεων που κάναμε πέρσι εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν θα είναι αποδυναμωμένη η στάση μας στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο γιατί πραγματικά ε, υιοθετεί μια πολύ πιο σύγχρονη στάση από ό,τι οι δύο αυτοί Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Άλλα μέλη τη Επιτροπή ΔΕΚ, ο κ. Βανίστελρο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα για μια επόμενη επταετία. Μπορεί κανείς να φιλοσοφήσει πολύ, αλλά είναι και πολύ ρεαλιστικό. Εμείς δίνουμε δίνουμε ε, τις, ε, τους προσανατολισμούς. Δείτε τι συνέβη στη διάρκεια της κρίσης. Ε, υπήρξαν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τις επενδύσεις και το, τα, τα, τα ταμεία βοήθησαν πολύ στην ανάκαμψη. Τώρα μιλάμε για τις περιφέρειες, για τις πόλεις. Όπως είπε ο Γιούνκερ, Θέλουμε να ξανασυνδέσουμε τους πολίτες με τα ευρωπαϊκά ιδανικά και όραμα. Είναι πάρα πολύ, καλό, πολύ σημαντικό να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Συνεχίζεται ένα εργαστήριο για τον προγραμματισμό, για τις περιφέρειες και το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε καλύτερα να το παρουσιάσουμε δεν είναι μόνο η αλλαγή των χρηματοδοτικών μέσων, ε, βεβαίως και αυτό, αλλά αυτό είναι, που είναι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια άλλη σχέση στην εταιρική σχέση και εκεί συμφωνώ απόλυτα με τους εισηγητές ότι ένας κώδικας διοντολογίας και η αρχή αυτή της εταιρική σχέσης θα πρέπει να μας βοηθήσει να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα και να υπάρχει μια ευθυγράμμιση. Όταν πηγαίνουμε με την Επιτροπή Ρέντζι, με τις αντιπροσωπείες μας, Είχαμε τρεις ε, φέτος και τρεις πέρσι και ακούει κανείς τους δημάρχους λένε ότι θέλουν να συνδέσουν στις πόλεις τους, στα χωριά τους και μπορεί να συζητήσουμε για το πώς θα γίνει αυτό. Και πολύ συχνά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό κομμάτι, να μην ξεχνάμε τις υποδομές. Ε, μπορούμε να δούμε λοιπόν πώς θα κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία αυτές τις ε, τους εκ των προτέρων όρους στην ακρόαση που κάνουμε εμείς στο ΕΛΚΑ υπάρχει κόσμος που έλεγε ότι στο δικό μας προγραμματισμό, ο δικός μας προγραμματισμός στα Υπουργεία, στις Περιφέρειες έχει βελτιωθεί και στα παλιά κρατημέλη και στα νέα κρατημέλη. Και γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε με τους στόχους κλειδιά που έχουμε στο, στο, στο ε, κανονισμό ήδη και να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε επανάσταση εδώ. Υπάρχει πίεση βέβαια στον προϋπολογισμό για τη συνοχή. Έχουμε λιγότερο 45% στο Ταμείο Συνοχής. Θα πρέπει να τα κάτι μελη να μπορούν καλύτερα να πούν πώς επιθυμούν να δαπανίσουν τα χρήματα. Αν έχεις λιγότερα χρήματα πρέπει να είσαι πιο κοντά στο πρόγραμμα του κράτους μέλους. Πρέπει να είσαι πιο κοντά στο προγραμματισμό της περιφέρειας και της πόλης και να τους δώσεις και περισσότερο λόγο. Αυτό εν μέρει το κάνουμε με τον κανονισμό Omnibus ήδη. Αλλά πρέπει να κάνουμε και ένα παραπάνω βήμα κατά τη γνώμη μου, να έχουμε πιο συγκεκριμένα μέσα, περισσότερη ευελιξία ίσως, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό θα το δούμε ίσως με τις τροπολογίες. Πάντως εν γέννη είμαι ευτυχής με αυτό που παρουσιάσατε γιατί είναι σταθερό, δεν δημιουργεί πολλά προβλήματα για τις περιφέρειες και τις πόλεις. Είναι σαφές καθοδηγείται από γνώση και από, με, το στόχος που έχουμε θέσει και στηρίζεται στα όσα είχαμε την περασμένη περίοδο. Ας μην χάσουμε χρόνο λοιπόν στην επόμενους μήνες και συμφωνώ με τη γνώμη της Κωνσταντσε ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε το Δεκέμβριο. θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω επιπλέον συνεδριάσεις για να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Ευχαριστώ η κυρία Μπρέσο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να παρέμβω για να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, όχι πολύ, αλλά λίγο παραπάνω χρόνο για την υποβολή τροπολογιών, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε με προσοχή την έκθεση και να προετοιμάσουμε τις ε, τροπολογίες μας. Αν είναι δυνατόν, λοιπόν, λίγο περισσότερο χρόνο. Θα θέλαμε. Πολύ θα χαιρόμασταν, τουλάχιστον εγώ πολύ θα χαιρόμουν. Τώρα, επί της ουσίας, εκτός ε, της, της ευχαριστίας μου προς τους δύο εισηγητές ε, που έκαναν ε, πολύτιμη δουλειά και πολλή δουλειά γιατί πρόκειται για έναν κανονισμό περίπλοκο. Ήθελα λοιπόν να παρέμβω για αυτό που έλεγε πριν ο συνάδελφος Ζουιτεμπουργκ. Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε μια πιο σύγχρονη στρατηγική και στην πολιτική συνοχή εν γέννη και στην πολιτική, ε, την επενδυτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως αφορά τους στόχους και από αυτού οι προτάσεις είναι ενδιαφέρουσες. Υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη συγκέντρωση, προσανατολιζόμαστε στους ε, κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους έχουμε άλλωστε συζητήσει όπως ας πούμε για τους ε, περιορισμούς στις εκπομπές. Άρα λοιπόν οι στόχοι των πολιτικών θα πρέπει να προσαρμόζονται και στους καιρούς. Μιλάμε για μια Ευρώπη μετά την κρίση που πρέπει να νοικοδομήσει εκ νέου την οικονομία της. Αυτό είναι ο κανονισμός που ορίζει τους κανόνες χρήσης των κονδυλίων. Επ' αυτού λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τελικά η καλή νόμη είναι η παλιοί νόμη. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι το να αλλάξει κανείς κανονισμό πάντοτε είναι θετικό, γιατί έχουμε να κάνουμε με κανονισμούς που αργά ή γρήγορα πρέπει να εφαρμοστούν από κράτη και περιφέρειες, αλλά και από τις τοπικές ε, αρχές, που είναι οι τελικοί χρήστες, και οι οποίοι προτιμούν να μην βλέπουν κάθε φορά αλλαγές στην δομή του κανονισμού. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου δεδομένο η μικρή αλλαγή δεν σημαίνει βέβαια ότι λείπουν οι καινοτομίε στην προγραμματική πρόταση. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν καινοτομίε και όχι τόσο στην αλλαγή των κανόνων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η σημαντική μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ένωσης είναι πολύ σοβαρή γιατί είναι αλήθεια ότι τα κράτη θα έπρεπε να αυξήσουν τη δέσμευσή τους στις επενδύσεις. Επ' αυτού δεν υπάρχει αμφιβολία, ωστόσο δεν έχουμε ακόμα βγει από την κρίση τελείως. Πολλές από τις χώρες και τις περιφέρειές μας δεν έχουν ε, βγει από την κρίση και έχουν δυσκολίες να ε, φτάσουν στο 50-60% στους ποσοστά χρηματοδότησης και να φτάσουν και στο 30% για τις πιο φτωχές περιφέρειες που είναι ακόμα πολύ φτωχές γιατί οι ανισότητες ε, στη διάρκεια της κρίσης αυξήθηκαν και δεν έχουν ακόμα βληθεί πολύ πολύ μερικός Γι' αυτό λοιπόν και πιστεύω ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί η επιλογή των ε, ε, των ε, εισηγητών μας να μην το καταστήσουν δέσμευση, υποχρέωση. Γιατί μετά δεν θα είναι εύκολη χρήση αυτών των πόρων. Και έπειτα, για τον ενιαίο κανονισμό, ακριβώς να πω ότι την περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε το αίτημα μιας ατζέντα για τις ε, ε, ε, περιοχές της Υπέθρου και τις ορεινές περιοχές και το θέμα τη ανάπτυξης πέθρου δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη γεωργία. Αυτό θα αποτελούσε βήμα προ τα πίσω. Οι περιοχές τη πέθρου θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλευτούν και οι ορεινέ περιοχές επίσης να εκμεταλλευτούν πλήρως τον προγραμματισμό αυτό που δεν είχε πάντα όλες τις τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να είχε επανειλημμένα στο πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού χρειάστηκε να βγει αυτό προς τα έξω, να γίνει δηλαδή ένα βήμα ε, που δεν θα πρέπει όμως να οθήσουμε και να πιέσουμε, γιατί ακριβώς ο προγραμματισμός δεν έχει πάντοτε απορροφηθεί πλήρως. Αυτό αυτός είναι ένας εξυγχρονισμός, ένας τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά με τις περιφερειακές πολιτικές και όχι να πάμε πίσω. Εγώ έχω κάποιες εμφιβολίες όπως ξέρει η κυρία Κρέλ αλλά όχι ο κύριος ε, σχετικά με την δυνατότητα να αφιερωθεί ένα μικρό κομμάτι των ε, προγραμμάτων συνοχής τα εθνικά τμήματα του Invest EU. Επειδή αυτό είναι εθελοντικό, γίνεται σε εθελοντική βάση και σε εθελοντική βάση εκ μέρους των περιφερειών, αν ε, είναι δυνατόν να εγγυηθούμε ότι αυτό θα γίνει με σεβασμό προς τη βούληση των περιφερειών, θεωρώ ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει αλλά είναι μια συζήτηση μόνο αυτή. Δεν έχω βεβαιότητες, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες απλώς ότι τα μόνα κονδύλια που συνδέονται με το InvestEU θα προέρχονται από τις ε, διαρθρωτικές ε, ε, πολιτικές, από τα διαρθρωτικά ταμεία, γιατί όλα τα άλλα, ε, και τα λοιπά, ε, συνδέονται ήδη. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι μάλλον θα είναι υπέρ ε, των διαρθρωτικών και των περιφερειακών πολιτικών. Για τα κοινωνικά ε, κονδύλια, παραδείγματο χάρη, είναι οι επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές θα μπορούσαν να ευνοήσουν ε, νέες μορφές του InvestEU που δεν θα είναι πια το κλασικό σχέδιο Juncker. Θα έχουν άλλες βασικές αρχές στο προγραμματισμό τους. Αυτά, αλλά ομολογώ ότι δεν έχω ακόμα αρκετά κατασταλαγμένες απόψεις, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες πάνω στο σημείο αυτό της πρότασης. Ε, για όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή, μια εξαιρετική βάση ε, για τις εργασίες μας και τις ε, συζητήσεις μας και ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να επιδείξει μεγάλο θάρρος γιατί ε, συζητείται πολύ η πολιτική συνοχή στα τελευταία χρόνια ε, δέχεται πολλές επιθέσεις ενώ ε, από την άλλη πλευρά εγώ θεωρώ ότι είναι η πιο αποτελεσματική πολιτική η πιο σημαντική πολιτική ε, εξισορρόπησης των περιφερειών και υποστήριξης της ανάπτυξης των πιο των λιγότερων επιτυμένων περιφερειών πιστεύω ότι είναι σε θέση η πολιτική αυτή να δώσει μια νέα όθηση. Είναι, ε, θα πρέπει να παραμείνει ένας πυλώνας της πολιτικής μας και θα πρέπει να την υπερασπιστούμε και σε οικονομικό επίπεδο με όλες τις δυνάμεις μας. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορώ να συμφωνήσω ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν τα αντίστοιχα ποσά σύμφωνα με τις προτάσεις που θα κάνει το Κοινοβούλιο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ο κύριος Σέρτμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους ε, συνεισηγητές για τη σκληρή τους δουλειά. Και πράγματι νομίζω πως ε, έχουν επιτύχει πολλά θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Το δεύτερο τώρα είναι ότι συμφωνώ και εγώ ότι χρειαζόμαστε σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική συνοχή σήμερα περαιτέρω εξέλιξη, όχι επανάσταση σε ό,τι αφορά την άσκηση αυτή της πολιτικής. Γιατί όπω ακούστηκε σήμερα στην ε, αίθουσα παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν την αξιοποίηση αυτών των κοντιλίων, όχι μόνο κατά τελευταία χρόνια αλλά και γενικότερα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε εξέλιξη εδώ και όχι επανάσταση, γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει όταν προσπαθούμε να βάλουμε μια επανάσταση. Ε, και συμφωνώ λοιπόν με αυτά που προτείνουν εδώ οι συγκητέ ε, και ε, οι ταχύς ρυθμοί με τους οποίους εργάζονται οι συγκητέ σε αντίθεση με άλλες μας εκθέσεις είναι πραγματικά κάτι το ευπρόσδεκτο και για τους τελικούς δικαιούχους αυτών των κοντιλίων που θα ωφεληθούν από αυτά τα κοντιλία. Γιατί όσο πιο γρήγορα υιοθετήσουμε τους κανόνες και τις αλλαγές που θα επιβάλλουμε σε αυτούς τους κανόνες σε ό,τι αφορά αυτά τα ταμεία, τόσο πιο νωρίς οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν και θα γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτά τα κονδύλια και έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν και τα μικρότερα project στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα έλεγα ότι είναι προτιμότερο να έχουμε ένα κείμενο το οποίο ναι δεν είναι τέλειο, αλλά μπορεί να αποτελέσει καλή βάση εργασία, ένα κείμενο πάνω στο οποίο μπορούν να εργαστούν οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με το να ε, καθυστερήσουμε για μήνε, σε ό,τι αφορά αυτό το ε, κείμενο, ε, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε και στο να περάσει, για παράδειγμα, το νέο κοινοβούλιο στο να ξεκινήσει μια συζήτηση ω προ το αν είναι καλό πράγμα ή όχι, πολιτική συνοχή και ούτω καθεξής. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τι περιοχε 1 NSYN2 σε σύγκριση με τις 1 3 ε, νομίζω, και αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι ε, δεν είναι ε, εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε. Γιατί το 1 3 είναι πιο χρήσιμο, ειδικότερα στην περίπτωση μακροπρόθεσμων μεγάλων έργων τα οποία συνεπάγονται και υψηλά σε υψηλό κόστος. και αυτό αφορά ειδικότερα τη τελευταία φάση της ε, υλοποίησής τους. Ε, ταυτόχρονα το N2 μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμετα αποτελέσματα όπως ε, για παράδειγμα στην πλασματική αν θέλετε κατανομή, το σπάσιμο αν θέλετε το project σε μικρότερα κομμάτια ακριβώς επειδή οι χρονικοί ορίζοντες για αυτά τα project είναι πλέον μικρότεροι. Επίσης με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βάλουμε ένα φραγμό στην καινοτομία γιατί τα καινοτόμα έργα συνήθως απαιτούν περισσότερο χρόνο για την υλοποίησή τους έτσι ώστε δηλαδή να επιτευχθούν ακριβώς αυτά τα μεγάλης σε αποτελέσματα της καινοτομίας σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Αυτά, λοιπόν, αυτός ο αντίκτυπος της καινοτομίας ε, συχνά δεν μπορεί να επιτευχθεί. Κάτι ακόμα που αναφέρθηκε είναι αυτή η μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης ε, από 85% σε 70% σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Και εδώ και πάλι να πω ότι εάν ο στόχος εδώ ήταν να αναλυθούν περισσότερες ευθύνε από την πλευρά των κρατών μελών ακριβώς μέσω τη αύξηση του σχετικού ποσοστού συγχρηματοδότηση που βαρύνει τα κράτη-μέλη, τότε θα πρέπει να σας πω ότι μάλλον θα απογοητευτείτε. Ε, αν αυτή είναι πραγματικά η πρόθεση, τα πράγματα δεν νομίζω πως θα εξελιχθούν με τον τρόπο που νομίζετε, γιατί στην πράξη αυτή η συγχρηματοδότηση μειώνεται ακόμα περισσότερο μέσω άλλων ε, κανόνων και κανονισμών ε, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τις ε, προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την ε, συγχρηματοδότηση. χρηματοδότηση. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά σήμερα το ποσοστό στη χρηματοδότηση είναι 85%, στην πραγματικότητα σήμερα βρίσκεται στο 64%. Αν λοιπόν τώρα προβλέψουμε στο νόμο 70% ουσιαστικά στη χρηματοδότηση θα μειωθεί σε λίγο παραπάνω από 50%. Και αυτό τι σημαίνει με τη σειρά του ότι θα υπάρξει ένα φράγμα χρηματοδότησης για project σε διάφορες ε, περιοχές. Επίσης, Νομίζω πως θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης των χρηματοδοτικών εργαλείων, γιατί εδώ υπάρχει τεράστιο ε, δυναμικό για το μέλλον. Συνοψίζοντας, για να ολοκληρώσω, να πω ότι είναι καλύτερο να ε, συμφωνήσουμε επί ενός εγγράφου, το οποίο δεν θα είναι τέλειο, αλλά να το έχουμε έγκαιρα στη διάθεσή μας, προκειμένου να το έχουν έγκαιρα στη διάθεσή τους όλοι όσοι είναι ενδιαφέρονται για αυτά τα κονδύλια. Και βέβαια αυτό το ε, σύστημα που θα προβλέπει θα είναι ε, το, όσο το, πιο, το δυνατόν πιο απλό Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι πραγματικά, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο αυτό το έγγραφο και τέλειο ο κανονισμό, θα ε, επιτύχει τα σωστά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο, ο κύριο Όλμπριχτ. Θα ήθελα να στήσω συγγνώμη γιατί τα όσα θα πω ουσιαστικά ήδη υπόθηκαν. Απλώ θα ήθελα να ευχαριστήσω του ε, συνσηγητέ, ε, αλλά όχι συμβολικά, αν θέλετε, γιατί πάντοτε του ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ πραγματικά γιατί βρίσκονται, αντιμέτωποι με μια νέα πρόκληση. Δηλαδή, ε, καλούνται να τοποθετηθούν σε μια περίοδο όπου βρίσκεται αναθεώρηση σχετική ε, πολιτική. Ε, δηλαδή δεν είναι εδώ μια συνήθι διαδικασία. Εδώ είναι τελείω διαφορετική η πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Και με κάθε σεβασμό απέναντι στον συνάδελφο να πω ότι δεν συμφωνώ αυτό που είπε ότι το Συμβούλιο είναι πιο μοντέρνο στην τοποθέτησή του. Ε, και αυτό γιατί, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων στο ίδιο το Συμβούλιο. Υπάρχουν δηλαδή κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο που θεωρούν ότι ο μόνος τρόπος, η μόνη ευκαιρία που έχουν για να εξυγχρονιστούν, για να επιτύχουν καινοτομία είναι μέσω της πολιτικής συνοχής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, η μόνη τους ευκαιρία είναι η πολιτική συνοχής. Ενώ άλλα κράτη-μέλη όπως για παράδειγμα οι κάτω χώρες, η Δανία, η Σουηδία, δεν επιθυμούν κανένα είδου πολιτική συνοχή. Και θέλουν λοιπόν αυτή η πολιτική συνοχή να κατευθυνθεί ως υποστήριξη συνοχή προ τι φτωχότερε χώρε. Και σα το λέω αυτό γιατί είχα μια συνάντηση με του ε, πρέσβει από αυτέ τι χώρε οι οποίοι μου είπαν, εγώ σε μένα ως εισηγητή για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ότι η καλύτερη λύση για εκείνους είναι 0% κόστος για του φορολογούμενου σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Ουσιαστικά δηλαδή μου είπαν ότι δεν χρειαζόμαστε πολιτική συνοχή. Εντάξει, αυτή είναι επίσημη θέση του, τελικά μπορεί να είναι διαφορετική. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ανεπτυγμένε χώρε δεν χρειάζονται πολιτική συνοχή. Ενώ ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να κατευθύνεται στι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Ενώ η πρόταση τη Επιτροπή τώρα είναι τελείω διαφορετική. Είναι αντίθετη. Ουσιαστικά λέει πολιτική συνοχή για όλου και προκειμένου να είναι διαθέσιμη για όλου ε, προβλέπει διαφορετικά κριτήρια. Γι' αυτό ε, έγινε και αυτή η αναφορά σε ό,τι αφορά αυτέ τι μεταβατικέ ε, περιοχέ. Ακριβώ γίνεται αυτή η διαφορά, η αλλαγή στην φιλοσοφία. Αυτή λοιπόν είναι η νέα πρόταση τη Επιτροπή ότι πολιτική συνοχή θα πρέπει να ισχύει ε, για όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, για τα φτωχότερα ενδεχομένω λίγο περισσότερη υποστήριξη, για τις ε, περιοχέ τι μεταβατικέ κάπως λιγότερη, αλλά πολιτική, δηλαδή υποστήριξη σε επίπεδο πολιτικής συνοχής για όλους. Και όταν ακούμε τα όσα λένε η Επιτροπή και το Συμβούλιο, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι η ειδική μεταχείριση, η προνομιακή μεταχείριση των νέων κρατών μελών ε, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Άρα λοιπόν αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μα. μας. Ε. Ότι δηλαδή πάμε πλέον αυτή η δική μεταχείριση, καλύτερη μεταχείριση των νέων κρατών μελών. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξή. Άρα λοιπόν ε, το... Εκείνο που μπορεί να συμβεί ο κίνδυνο είναι αυτέ οι χώρε, οι οποίε δηλαδή συμβάλλουν περισσότερο στον προπολογισμό, ε, να πιέσουν τελικά στο να οδηγηθούμε σε μια παραδοσιακή πολιτική συνοχή θα λένε ουσιαστικά ότι με τα υπόλοιπα κονδύλια μπορούμε ακριβώ να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινοτομία και το καθεξή. Και αυτό είναι ο κίνδυνο βέβαια να συμβεί κάτι τέτοιο. Και γιατί είναι ο κίνδυνο, Γιατί ο, η ιδιαιτερότητα τη πολιτική συνοχή δεν είναι τα χρήματα, είναι η κοινή διαχείριση. Η κοινή διαχείριση είναι τελικά που έχει αποφασιστική σημασία. Η συνευθύνη, η κοινή ανάληψη ευθύνη, η κοινή συγχρηματοδότηση που είναι κλειδί για την πολιτική συνοχή. Είναι η συνολική διαχείριση τη όλη πολιτική και η άσκηση επιρροή ε, των κρατών μελών στη λειτουργία αυτή τη πολιτική συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν όταν ε, συζητήσαμε τον κανονισμό για τις γενικές διατάξεις ε, και αναφέρθηκε αυτή η, το, το, να φύγουν αυτά τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής ουσιαστικά αναφερόταν η, το να φύγουν αυτά τα κονδύλια από την κοινή διαχείριση γιατί αν τα πάρουμε αυτά τα κονδύλια από τους σχετικούς φακέλους και τα βάλουμε για παράδειγμα στους εθνικούς φακέλους για παράδειγμα στο ΣΕΠ Δηλαδή, πάρουμε αυτά τα κονδύλια ουσιαστικά από την κοινή διαχείριση και τα μεταβάσουμε στου εθνικού φακελούς στην εθνική διαχείριση. Ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Μειώνουμε τα κονδύλια τη πολιτική συνοχή. Και αυτή είναι η τάση. Το ίδιο συμβαίνει και στο επίπεδο του InvestEU. Δεν θέλω να πω ότι είναι κακή ιδέα το InvestEU, αλλά γιατί έχει εθελοντικό χαρακτήρα το InvestEU γιατί όλοι θα προσπαθήσουν να επιλέξουν τον τρόπο ο οποίο είναι ευκολότερο για εκείνους. Το InvestEU θα είναι ευκολότερο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Γιατί λοιπόν να μην καταστήσουμε πιο απλή την πολιτική συνοχή από το να μεταβιβάζουμε τέτοια κονδύλια σε ένα πιο απλό σύστημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Το αν θέλουμε να διατηρήσουμε λοιπόν μια τέτοια είδους, ε, μια τέτοια πολιτική η οποία δεν είναι περιοδοσιακή και δεν με αυτόν τον τρόπο δεν είναι παραδοσιακή, αλλά βασίζεται στην κοινή διαχείριση. Θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα δηλαδή. Θα υπάρχει κοινή διαχείριση ή όχι αυτή τη πολιτική. Και από εκεί μετά σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Θέλετε αυτό το περιεχόμενο και ε, κατευθύνεται και εστιάζει περισσότερο στην καινοτομία ή όχι. Για παράδειγμα, οι γύρω συντη μα είπαν ότι δεν θεωρούν πως θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η έρευνα από τα δικά του κονδύλια. Δεν, τους, δεν τις αφορά θα μπορούσε η συνοχή δηλαδή να αφορά τη διαχείριση την αστική σε ό,τι αφορά την κοινοτομία, για παράδειγμα στι μεταφορέ ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι το πρόβλημα και θα γίνει κάποια συζήτηση σε σχέση με αυτό το ζήτημα, δηλαδή τη μεταφορά κάποιων κονδυλίων από τα ε, ταμεία στον, ε, στο ΣΕΦ, στην, στο Μηχανισμό Συνδέοντα στην Ευρώπη και από εκεί και μετά τι θα γίνει και σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση αυτού των κονδυλίων στο InvestEU. Εδώ επαναλαμβάνω αυτό που έχω ήδη πει σε αυτή την Επιτροπή. Ε, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αυτή η μεταβίωση ό,τι αφορά του εθνικού φακέλου στο InvestEU χωρίς ε, την, ε, την, το, το κοινοτικό κομμάτι, το ενωσιακό αν θέλετε κομμάτι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει, υπάρξει πλήρης κατακαιρματισμός αυτών των κονδυλίων μέσα στο InvestEU. Συνοψίζοντας, λοιπόν να πω ότι θεωρώ ο κανονισμό ε, CPR αποτελεί ένα πολύ βασικό έγγραφο ε, και στην έκθεσή μας θα τοποθετηθούμε ως προς το κατά πόσο συμφωνούμε με αυτή τη νέα γραμμή που ακολουθεί η Επιτροπή ή όχι. Και νομίζω πως ε, ο κ. Σάκη μας σωστά το ανέφερε ότι δηλαδή το ε, ο στόχο μα δεν είναι εδώ να δημιουργήσουμε μια νέα επανάσταση. Αλλά νομίζω πως δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια τέτοια δύσκολη συζήτηση. Ε, γιατί βέβαια το ζητούμε εδώ δεν είναι να βρούμε μια λύση γρήγορα, είναι να φτάσουμε σε μια ε, θέση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όρους εδώ στην ε, πολιτική ρέτζη όπως παλιά πολιτική, παραδοσιακή πολιτική, γιατί με αυτό το, το,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 Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη επειδή έφτασα αργοπορημένος λόγω άλλων υποχρεώσεων που είχα εδώ σε αυτό το κτίριο. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συνεισηγητές για την εργασία τους. Έχουν αντιμετωπίσει αντιμετωπίσουν μεγάλη πρόκληση για να βρουν συμβιβαστικές λύσεις όσον αφορά το επόμενο, τις επόμενες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με την πολιτική συνοχής. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τους δύο πολύ για την εργασία σας και να εκτιμώ ποια είναι η εκτίμησή μου για την πρόταση της Κομισιόν, διότι είμαι βέβαιος ότι θα ε, προσφέρει μεγαλύτερη απλούστευση και ε, ομοιομορφία στους κανόνες. Όμως, είναι αρκετά φιλική προς το, φιλικός μάλλον προς το χρήστη αυτός ο κανονισμός. Προσπαθούμε να επιτύχουμε ωφέλη για τους δικαιούχους, για τους χρήστες αυτής της κατευθυντήριας γραμμής και του κανονισμού. και να καταργήσουμε άχρηστες ε, διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις προηγούμενες, ε, στο προηγούμενο κανονισμό. Για τις περιοχές της υπαίθρου που πολλές φορές είναι η σταχτοπούτα των ε, κανονισμών. Χρειαζόμαστε περισσότερες απλοποιήσεις και πιο αποτελεσματικά μέτρα ώστε να μην ε, απεριμωθούν περισσότερο οι ερηνές και οι γεωργικές περιοχές. Γι' αυτό το λόγο οι κανόνες θα πρέπει να είναι όσο γίνεται απλούστεροι. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που συνορεύει με τη Σλοβακία και δις εξελέγει δήμαρχος ενός μικρού δήμου. Γι' αυτό θα, ε, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την, την πολιτική συνοχή με την πολιτική γεωργία. Γι' αυτό θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Επιτροπή. Οι συγκητέ έχουν να παίξουν πολύ σπουδαίο ρόλο να πιέσουν την Κομισιόν ώστε να λάβει ακόμη πιο απλά μέτρα να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα έπειτα για την ε, ε, χρηματοδοτική για, τις, ε, τα κονδύλια, τα χρηματοδοτικά. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που προτείνεται μπορεί να αποθαρρύνουν πολλούς δικαιούχους από το να ε, χρησιμοποιήσουν ε, τα κονδύλια. Και αυτό έχει να κάνει και με τους κανόνες 1 2 και 1 3. Στην Τσεχία τι θα μπορούσε να συμβεί ότι το έτος ανάπτυξης θα είναι ένα μόνο. Η τρέχουσα περίοδος θα ολοκληρωθεί στον νησιν 3 και η επόμενη περίοδος στο νησιν 2. Άρα λοιπόν μέχρι τότε σε ένα χρόνο θα πρέπει να απορροφηθούν αυτά τα κονδύλια. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Τσεχία, αλλά και την Πολωνία, τη Σλοβακία και άλλες χώρες. Δεν θα έχουμε δηλαδή το διοικητικό μηχανισμό για να ε, ε, σχεδιάσουμε ολοκληρωμένα προγράμματα. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε μια μεταβατική περίοδο πριν την έναρξη, ώστε το νη συν 3 να αρχίσει στην αρχή, να ισχύσει μάλλον στην αρχή της νέας προγραμματικής περίοδου. Τελευταίο μου σχόλιο. Επικρατεί μια περίπλοκη κατάσταση στην αγορά εργασία. Διάφοροι εργα... Ε, εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και καθόλου στον δημόσιο ή στον ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασχολούνται με ιδιωτικά project. Αυτή λοιπόν η συγκέντρωση στις αρχές της νέας προγραμματικής περίοδου μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση όπου δεν θα έχουμε αρκετά το κόσμο για να ε, φτιάχνει νέα project. Σίγουρα αυτό θα συμβεί σε διάφορα κρατημέλη, αλλά εκεί που υπάρχει κάτω από 5% απασχόληση, εκεί θα λείψουν οι διοικητικές δυνατότητες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αυτή, αυτό ήταν το, ε, η τελευταία παρέμβαση από τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι τώρα θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Χαβιέρτο Σορίτ, που είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Θα μιλήσω την Ισπανική. Ναι. Για να σας πω καταρχάς ε, πολλά ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας επιτρέψει να εκθέσουμε τις ε, απόψεις της Επιτροπής μας σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και επίσης γενικότερα για τη συνεργασία ε, γιατί για πολλά θέματα στα οποία, ε, τα οποία μας απασχολούν εδώ στο Κοινοβούλιο όπως και στην Επιτροπή μας τις επόμενες ε, φάσεις έχουμε έρθει σε επαφή με τους εισηγητές, πράγμα το οποίο μας οδηγεί πιο εύκολα στο να συντάξουμε καλές ε, και συντονισμένες εκθέσεις. Εγώ είμαι εισηγητής ε, και, ε, για τον Γενικό Κανονισμό και αντικαθιστώ εδώ τον Στέφανο Μάλια που είναι ε, ε, μαλλιά που είναι ε, επιχειρηματίας και το λέω γιατί υπάρχει μεγάλη συνένεση στην ψηφοφορία των κειμένων μας και στους από τους τρεις τομείς της Επιτροπής μας, δηλαδή και από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες και από τους ε, διοικητικούς υπαλλήλους. Ξεκινήσαμε ε, λοιπόν να συζητάμε για την ε, με, την ανησυχία για τις περικοπές ε, που γίνονται ενώ σοβεί ακόμα η κρίση σε πάρα πολλές χώρες και τώρα διαπιστώνουμε και ζούμε τις πολιτικές συνέπειες ε, και τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης ότι δηλαδή ε, φαίνονται πολιτικές τάσεις οι οποίες αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν νέα project τα οποία μπορεί να στηρίξουν την εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα ε, βλέπουμε ότι αυτές οι περικοπές ε, δημιουργούν, προκαλούν μεγάλες δυσκολίες. Άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι ότι ε, αυτό το deficit που έχουμε, το έλλειμμα που έχουμε, είναι το έλλειμμα στις επενδύσεις μεταφορά από κονδυλίων από δεξιά στα αριστερά. Το θέμα είναι ότι το σύνολο των κονδυλίων των ευρωπαϊκών θα σημαίνει μείωση των επενδύσεων. Ενώ αντίθετα αυτό που χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο είναι περισσότερες επενδύσεις. Εν πάση περιπτώσει η μεταφορά κονδυλίων για να συμπληρωθεί ένα project ε, επενδυτικό έχει νόημα με αυτό το invest away, αλλά αυτό που θα είχε μεγαλύτερο νόημα ήταν να μην υπάρχουν και περικοπές. Εν γέννη, συμφωνούμε με τις προτάσεις του Κομισιόν που θέλει να αυξήσει το συνολικό ποσό των ε, εσόδων και των δαπανών ε, στο 3% του ε, καθάριστου εγχωρίου προϊόντος και να παραμείνουμε δηλαδή στα επίπεδα που είναι αντίστοιχα με το τρέχον πλαίσιο, δηλαδή το 2014 με 2020. Συμφωνούμε με τα όσα υπόθηκαν εδώ για τις τροποποιήσεις που ενισχύουν την απλούστευση, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα. Συμφωνούμε βεβαίως ε, για ορισμένα επίπεδα ενίσχυσης ε, της ε, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όμως θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε ένα στοιχείο το οποίο αναφέρεται στον κώδικα διοντολογίας. Υπάρχει δηλαδή εκεί μια σοβαρή αντίρρηση του Business Europe και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εδικάτων όσον αφορά το συγκεκριμένο κώδικα. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή και συζήτηση των οργανώσεων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έπρεπε να ζητήσουμε λοιπόν από την Κομισιόν να προτείνει μια αναλλαγή ε, για έναν κώδικα διοντολογίας ο οποίος να είναι ε, δεσμευτικός. Ε, για τις ε, τροποποίησεις έχουμε ε, κάποιες παρατηρήσεις να κάνουμε με βάση την θέση της Επιτροπής μας. Δεν συμφωνούμε με τους μακροοικονομικούς όρους για να μπορέσουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια και μάλιστα με όσον αφορά την αυστηρή και άκαμπτη ερμηνεία αυτών των όρων. Συμφωνούμε για την αλλαγή από 2 στα 3 χρόνια την περίοδο εκτέλεσης, να περάσουμε δηλαδή στο συν 3 αντί για το συν 2 και όσον αφορά την συγχρηματοδότηση θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει μια πιο ευελικτή ε, θέση Ιδιαίτερα όσον περνάει κανείς από τις περιοχές σύγκλησης στις περιοχές μετάβασης που μπορεί να είναι ένα πολύ απότομο άλμα για πολλές χώρες. Θεωρούμε πως εκεί πρέπει να επανεξεταστεί. Επίσης όσον αφορά συγκεκριμένα μέσα για τις μειονεκτούσες περιοχές, με τα διευθυντικά προβλήματα τα μόνιμα, ας πούμε, ε, νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές, ε, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και να ενταχθεί και το Γεωργικό Ταμείο σε αυτές τις διατάξεις και δύο παρατηρήσεις ε, τελειώνοντας αφορούν το ότι διαφορούμε, διαφωνούμε γιατί διαγράφει από το άρθρο 7, εκεί που γίνεται λόγος για τους όρους για τις συμφωνίες, αφαιρέθηκαν όλες οι αναφορές που υπήρχαν στον ισχύοντα κανονισμό για την ε, πρόθεση της ισότητας ανδρών γυναικών, ε, τη την ε, απαγόρευση διακρίσεων. Ναι, είναι το 67 του κανονισμού. Ε, του ισχύοντος κανονισμού είναι σημαντικό αυτό λοιπόν που, άρθρο που αφορά τις εθνικές δεσμεύσεις για τις συμφωνίες ε, σύνδεσης κτλ να γίνεται η σχετική αναφορά ώστε να ε, είναι σύμμορφη, ε, σύμμορφος αυτός ο κανονισμός προς τους υπόλοιπους. Να τονίσουμε επίσης ότι στο πλαίσιο μιας τόσο μεγάλης ε, μείωσης των κονδυλίων θα πρέπει να είμαστε κατά της μεταφοράς προς τη διευκόλυνση ιδέοντας στην Ευρώπη. Όχι γιατί διαφέρουμε στο να, τον στο τονωθεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά γιατί είμαστε κατά της περικοπής γενικότερα. Να μεταφέρουμε ναι, στο InvestWay κάποιο κομμάτι των κονδυλίων που είναι στο Ταμείο Συνοχής, ναι, εκεί θα υπάρχουν προβλήματα. Δεν πρόκειται λοιπόν για α, α, αντίρρηση. Εξαρτάται, κανείς, εξαρτάται βεβαίως από το πώς ε, έχουν γενικότερα οι πολιτικές συνοχής και τη γενική χρηματοδότηση για τη συνοχή. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμο για μας που ακούσαμε την ε, άποψή σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε και ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Δυστυχώς η κυρία Μαρίνη, εκπρόσωπος της Επιτροπής των Περιφερειών, δεν μπόρεσε να ε, προσαρμόσει το πρόγραμμά της και να παρευρεθεί στη συνάντησή μας. Και έτσι τώρα θα συνεχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Φανπρέσκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους δύο εισηγητές για την απίστευτα πολλή δουλειά αυτή που κάναν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πραγματικά, όπως τονίστηκε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ε, ασφάλεια δικαίου για ε, τους δικαιούχους, ώστε να μην έχουμε ε, το πρόβλημα των καθυστερήσεων που αντιμετωπίσαμε και κατά την τρέχουσα περίοδο. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι κοινό στόχος αυτός της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζουμε την εστίαση της έκθεσης σε έναν επιλεγμένο αριθμό θεμάτων που υποτίθεται θα πρέπει να αλλάξουν, πράγμα στο οποίο δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά θεωρούμε ότι είναι μια καλή προσέγγιση αυτή και ελπίζουμε ότι στις συζητήσεις ε, που θα γίνουν στο Κοινοβούλιο θα επικρατήσει και εκεί αυτή η προσέγγιση. Γιατί αν γίνουν υπερβολικά πολλές αλλαγές επιτάπητος, ε, σίγουρα αυτό δεν θα είναι προς όφελος μιας ε, ταχείας προόδου των διαπραγματεύσεων. Μια άλλη γενική παρατήρηση. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την υποστήριξή μου προς την προσέγγιση που ε, επιλέγει για την έκθεση να μην αποδυναμωθούν, τονίζω να μην αποδυναμωθούν οι διατάξεις της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε ένα σημαντικό ρυθμό απλοποίησεων για να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος, αλλά δεν θεωρούμε ότι όλες αυτές οι απαιτήσει είναι περιττές. Θεωρούμε ότι κάποιες είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η λογοδοσία και η διαφάνεια, γιατί είναι χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών και ε, χαιρόμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζε την Κομισιόν στην προσπάθεια αυτή, γιατί ξέρετε ότι ε, ακούγονται προτάσεις να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρόταση απλοποίηση ε, για να προχωρήσουμε ακόμα πιο πολύ. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι τα χρήματα δεν θα πρέπει να δίνονται έτσι ε, δωρεάν, ας πούμε. Και γι' αυτό σε ευχαριστούμε για την προσέγγιση αυτή που υιοθετήσατε. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω σε τρία-τέσσερα από τα θέματα που θύχτηκαν κατά τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα οι οικονομικέ μεταρρυθμίσει και οι επενδύσει που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Πραγματικά θέλουμε να πλησιάσουν περισσότερο αυτές οι δύο διεργασίες. Και νομίζουμε, όπως είπε ο κύριος Όλμπερτ, ότι η επιμερισμένη διαχείριση, ο τρόπος δηλαδή αυτός ε, κατανομής των πόρων μας είναι μια μοναδική ε, ευκαιρία γιατί μας ε, ε, ε διευκολύνει να δημιουργήσουμε την έννοια του ownership σε όλα τα επίπεδα, και στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις. Επίσης θεωρούμε ότι αυτό μας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο να έχουμε μεγαλύτερη έμφαση και εστίαση στην περιφερειακή διάσταση, γιατί έχει παραμεληθεί μέχρι τώρα και επίσης μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και όχι μόνο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό θεωρούμε ότι βοηθάει να έρθει η πολιτική συνοχή πιο κοντά στο επίκεντρο της ε, δημοσιονομικής διακυβέρνησης που δεν μπορεί παρά να βοηθήσει μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω είναι το InvestEU. Πολλά επιχειρήματα ακούστηκαν, αλλά εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε ένα-δύο σημεία ε, τα οποία θέλω να υπογραμμίσω. Δεν πρόκειται για μεταφορά κονδυλίων, πρόκειται για συνεισφορά για να επιτευχθούν οι στόχοι της συνοχής. Αυτό συγκεκριμένα τι σημαίνει. Ότι το κράτος μέλος που σε εθελοντική βάση συνεισφέρει στο InvestEU θα υπογράψει μία συμφωνία συνεισφοράς όπου θα ορίζονται οι όροι και οι στόχοι για την χρήση αυτών των πόρων. Παράδειγμα, αν το κράτος μέλος θέλει τα χρήματα να κατανεμηθούν με βάση μια συγκεκριμένη κλίδα ε, κατανομής σε όλες τις περιφέρειες του ελόγω κράτους μέλους, φυσικά ο εταίρος που θα είναι είτε η Τράπεζα Επενδύσεων ή οποιοδήποτε άλλος εταίρος, θα πρέπει να σεβαστεί ε, τον τρόπο αυτό υλοποίησης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση παρέχει πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την κάλυψη κινδύνων, τη μόχλευση, τον διοικητικό φόρτο, αλλά και ε, μεγαλύτερο ποσοστό ε, οικονομιών κλίμακος. Αν δεν αποδώσει, αν ο εταίρος δεν μπορέσει να ε, ε ανταποκριθεί, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει πίσω τα χρήματα. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι μια εναλλακτική που είναι χρήσιμο να την έχουμε. Κανεί δεν σα υποχρεώνει να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά δεν πρόκειται για μεταφορά. Πρόκειται για επίτευξη των στόχων τη ε, πολιτική συνοχή μέσω διαφορετικών οδών. Δεν πρόκειται για μεταφορά κονδυλίων. Για το Ταμείο αγροτική ανάπτυξη. Εδώ ξέρετε ότι η Κομισιόν πρότεινε μια μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, που θα φέρει πιο κοντά τα δύο γεωργικά ταμεία, το ένα στο άλλο και πίσω από αυτή τη μεταρρύθμιση υπάρχει ε, ένα νέο μοντέλο όπου βασικά σύμφωνα με την κοινή γεωργική πολιτική θα απομακρυνθούμε από την συμμόρφωση ε, σε μια προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα. Και για να το επιτύχουμε αυτό, η Κομισιόν έκανε την πολιτική επιλογή που λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα και να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αν οι κανόνες που διέπουν αυτά τα δύο ταμεία θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Καταλαβαίνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαφορετική άποψη, αλλά απλώ θέλω να σα εξηγήσω έτσι γιατί ε, έχουμε καταλήξει σε αυτή την πρόταση. Δύο λόγια τώρα ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, για τον κώδικα δεοντολογίας. Ο κώδικας δεοντολογίας που εφαρμόζεται σήμερα ίσως δεν είναι τέλειος. Συμφωνούμε. Πέραν αυτού όμως υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο είπαμε ότι δεν θέλουμε να ανακαλέσουμε τον ισχύοντα κανονισμό και θέλουμε να συνεχίσει να ισχύει ο κώδικας διοντολογίας. Γιατί, Γιατί θέλουμε αυτή η εταιρική σχέση που ορίζεται πώς υποτίθεται θα πρέπει να δουλέψει, θα πρέπει να υπάρχει ήδη όταν θα αρχίσουμε να συζητάμε με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες για την επόμενη γενιά έργων. Αυτό θα αρχίσει από την άνοιξη του 2019, σε 4-5 μήνες το αργότερο. Αν τώρα, αυτή τη στιγμή, απορρίψουμε, καταργήσουμε τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας και περιμένουμε να υιοθετήσουμε έναν άλλο κώδικα δεοντολογίας πιο καλά επεξεργασμένο, πιο προηγμένο, υψηλότερη ποιότητας, αν και θα πω ότι και ο τωρινό είναι καλή ποιότητα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τίποτα ενισχύ ε, που, θα, που να, να, να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν οποιοδήποτε κώδικα δεοντολογίας. Γιατί ο κώδικα διοντολογία θα ισχύσει από τη στιγμή που θα υιοθετηθεί η νομοθεσία. Και αυτό, α είμαστε ειλικρινεί, δεν θα γίνει μέσα σε τρει-τέσσερι μήνε. Γι' αυτό πήραμε την απόφαση να μην προτείνουμε νέο άρθρο για τον κώδικα διοντολογία, απλώ να συνεχίσουμε την ισχύ του υφιστάμενου άρθρου και να ξαναδούμε του κανόνε όταν ε, ξεκινήσει η διαδικασία προγραμματισμού. Τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το θέμα των μεγάλων έργων. Όπως ξέρετε, προτείναμε να καταργηθεί η έννοια αυτή. Θεωρούμε ότι όσον αφορά τα μεγάλα έργα μπορούμε να βασιστούμε περισσότερο στα εθνικά συστήματα. Ε, πέραν αυτού όμως, επίσης ενισχύσαμε τη θέση μας, στην πρότασή μας μάλλον, το ρόλο της Κομισιόν ε, όσον αφορά την παρακολούθηση ε, των κριτηρίων επιλογής των έργων. Ε, η Κομισιόν δηλαδή μπορεί να ζητήσει από την διαχειριστική αρχή να υποβάλει τα κριτήρια για την επιλογή των έργων ε, ε, πάνω στα οποία θα κάνουμε σχόλια τα οποία πρέπει να γίνουν σεβαστά από την Διαχειριστική Επιτροπή. Διατηρούμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Και τέλος έχουμε εισαγάγει μια νέα έννοια πράξεων στρατηγικής σημασίας που θα συμπεριληφθεί σε όλα τα έργα, γιατί τα μεγάλα έργα αφορούν μόνο, μην ξεχνάτε, τις μεταφορές και το περιβάλλον και μόνο ένα υποσύνολο των κρατών μελών. Εδώ υιοθετούμε μια προσέγγιση ευρύτερη, γιατί, ε, όπως είπα, σε όλα τα έργα θα πρέπει να προσδιορίζονται αυτές οι πράξεις ε, στρατηγικής σημασίας και η Επιτροπή Παρακολούθησης θα εξετάζει την ε, ε, φυσική και την διοικητική εξέλιξη ε, και αυτή είναι μια αρκετή εξασφάλιση για μας, ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε μια ξεχωριστή κατηγορία ε, μεγάλων έργων, την οποία προτείνουμε να καταργήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ε, για όλα τα σχόλια, όλες τις παρεμβάσεις. Και όλα αυτά δείχνουν ότι ε, οι μελλοντικέ συζητήσει για αυτό το θέμα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Η κυρία Κρέλα έχει το λόγο. Ναι, δεν θέλω να σχολιάσω όλες τις πανεβάσεις που έκαναν ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Νομίζω πως θα έχουμε τη δυνατότητα στις ε, πολυάριθμες ε, συναντήσεις με τους σκιώδους συζητητέ να τα συζητήσουμε, αλλά και εδώ στην Επιτροπή μας. Ένα σχόλιο μόνο θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο έκανε ο Γιάνν Όλμπριχτ. Και αυτό είναι το εξή. Πράγματι, σε ορισμένες περιπτώσεις η πολιτική συνοχή δεν είναι εύκολο πράγμα. Και αυτό γιατί έχουμε αποφασίσει συνειδητά ότι δεν πρόκειται για μια διαχείριση την οποία διοργανώνει η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια πολιτική η οποία ε, εφαρμόζεται, η οποία σκείται από κοινού με ε, τις περιφέρειες, με τις πόλεις, με τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής ερωτήκησης. Άρα λοιπόν παρόλο την κριτική που μπορεί κανείς να ασκήσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής, νομίζω πως αυτό που καταφέραμε δηλαδή να είναι πολιτική ε, συνοχής κάτι το αποτελεσματικό για όσους συμμετείχαν, πραγματικά ε, είναι γεγονός και πραγματικά μπορεί να λέμε ότι είναι μια παραδοσιακή προσέγγιση που ακολουθούμε, αλλά πραγματικά είναι κάτι ε, το οποίο τελικά φέρνει τα χρήματα, φέρνει τα κοντήλια στις περιφέρειες. Ενώ το InvestEU και εκείνη η απόσταση από την πλευρά του Προέδρου Γιούνκερ ότι δηλαδή για κάθε ένα ευρώ αυτού του κοντιλίου θα προσελκυστούν 17 ευρώ σε επενδύσεις ήταν κάτι το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν απλά marketing αυτού του ε, σχεδίου. Άρα λοιπόν σε μια περίοδο που καλούμαστε να σκεφτούμε το πώς θα οργανώσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη που ε, προσανατολίζεται στο μέλλον ε, σε ό,τι αφορά και το κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο και ταυτόχρονα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη ε, ε, από την πλευρά των πολιτών στις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω πως ε, πραγματικά αυτή η παλιωμοδίτικη εντό εισαγωγικών προσέγγιση ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή είναι πραγματικά πάρα πολύ επίκαιρη. Και γι' αυτό θεωρώ πως αυτή η ακρογωνιαία λύθη, αν θέλετε, της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να τους ε, γιατί αποτελούν δυνατότητες για να βιώσουν τελικά οι πολίτες μας οι οποίες ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το τι ακριβώς μπορεί να επιτευχθεί με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και φυσικά όταν κάνουμε τέτοιες ε, προτάσεις ότι δηλαδή το Ταμείο ε, αγροτικής ανάπτυξης θέλουμε να περιληφθεί και πάλι στον κανονισμό. Προφανώς το γνωρίζουμε εδώ ότι δεν πρόκειται για μια απόφαση η οποία θα ληφθεί από την δική μας Επιτροπή. Αλλά οι διαπραγματεύσεις τρέχουν. Δεν ε, συζητάμε εδώ χωρίς να βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργίας και θα δούμε και τελικά ποιοι κανόνες είναι καταλληλότεροι για 1-2 ή 1-3 ή το πώς θα διαμορφωθούν τελικά τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Όμως για τα N2 και N3 νομίζω πως έχουμε, μια, ε, έχουμε υποβάλει μια πολύ καλή πρόταση σε ό,τι αφορά και τη μεταβατική περίοδο και τις σχετικές διατάξεις και από εκεί και μετά θα πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου κυρίε και κύριοι συνάδελφοι το εξή. γιατί όλοι σας έχει εμπειρία σε αυτό το τομέα. Δεν ξεκινάει ένα κράτος μέλος τον σχεδιασμό των προγραμμάτων του σε ό,τι αφορά τη νέα περίοδο προγραμματισμού χωρίς να έχει ολοκληρώσει τα προηγούμενα του έργα. Οπότε πραγματικά για αυτόν τον λόγο σκεφτόμασταν κατά πόσο θα ήταν δύσκολο να οδηγηθούμε σε μια ρύθμιση με το συν Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ποσοστών συγχρηματοδότηση, θα συμφωνήσω με του συναδέλφου που θέλουν να το αυξήσουν, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σε αυτή την περίπτωση και τα κατάλληλα κονδύλια. Εάν θέλουμε δηλαδή πραγματικά να προβλέψουμε υψηλά ποσοστά συγχρηματοδότηση σε ό,τι αφορά και τι ιδιαιτερότητε κάθε επιμέρου ε, περιοχή, ε, τότε σημαίνει ότι λίγα θα είναι τα έργα τα οποία θα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με βάση τα δεδομένα κόντυλα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και αυτό το ζήτημα κατά νου όταν κάνουμε λόγο για τα ποσοστά συγχρηματοδότηση. Και εδώ βέβαια τίθεται και το εξή ζήτημα. Λέμε ότι θέλουμε μια πάρα πολύ αποτελεσματική πολιτική συνοχή και γι' αυτό το λόγο επιθυμούμε την συνεργασία με το InvestEU, με το Horizon Europe, με το LIFE, με, ε, με το Μηχανισμό Συνδέοντα στην Ευρώπη, αλλά όχι συνεργασία με τον τρόπο της μεταβίβασης των κοντιλίων. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τη συνεργασία μεταξύ αυτών των μηχανισμών. Και είναι αληθές αυτό που υπόθηκε, δηλαδή τα ανατολικά ευρωπαϊκά ε, κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία δηλαδή προσχώρησαν τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι δυνατότητα να λάβουν αυτά, αυτή την υποστήριξη. Θυμάμαι πως αυτή η συζήτηση ήταν πολύ σημαντική και στην Πολωνία, ότι δηλαδή θα πρέπει ακριβώς να είναι δυνατός ο συνδυασμός ε, των ε, κοντιλίων του ε, Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με ε, το σχέδιο Juncker. αυτή λοιπόν την προσέγγιση θα πρέπει να την υποστηρίξουμε και νομίζω με τις προτάσεις που κάνουμε στην έκθεσή μας ακριβώς ε, κινούμε σε αυτή την κατεύθυνση και έχουν νόημα αυτές τις προτάσεις μας τουλάχιστον κατά τη δική μας άποψη αλλά από εκεί και μετά θα δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια όσο δυνατόν πιο κοινή θέση από τη δική μας πλευρά εδώ στην Επιτροπή μας και σε τελική ανάλυση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος, ο κύριος Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω στα βουλγαρικά. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Όπως είπε η κυρία Κρέλ, προετοιμαστήκαμε πολύ, ε, ακούσαμε και πολλά ε, σχόλια. τα οποία σωστά παρουσίασαν την κατάσταση. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια από τα σχόλια. Μας ρωτήσατε κατά πόσο θα ήμασταν κατά της μεταφοράς στην ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Όχι, δε, καθόλου. Αυτό που επιθυμούμε είναι η αμοιβαιότητα. Εφόσον θέλ, πρέπει να μειώσουμε στο ίμιση τα κονδύλια για το Ταμείο Συνοχής, δεν υπάρχει λογική να διατηρήσουμε όλες τις άλλες μεταφορές. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή τη θέση που αντιστοιχεί στην πρόταση της Επιτροπής. Όσον αφορά την συγχρηματοδότηση, έγιναν σχόλια ότι υπάρχουν περιφέρειες που χρειάζονται περισσότερη συγχρηματοδότηση. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι την αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης, δηλαδή της σημερινής. Και αυτό πιστεύουμε πως ήταν το μέγιστο που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ολμπρέχτη για αυτά που είπε γιατί πιστεύω ότι αυτά που έχουμε καταφέρει σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σύμφωνα με την θέση του Κοινοβουλίου. Έγινε και μια ερώτηση σε σχέση με τα μεγάλα project όπου ο κύριος Χέκμαν Ορίζουμε ένα κατόφλι 100 εκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει πως ένα σχετικά μικρός αριθμός ε, προγραμμάτων θα επηρεαστούν από αυτό. Θέλουμε όμως να τα, καλύψουμε, και να εξασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή τους, καθώς πρόκειται για πολύ ε, σημαντικά προγράμματα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βουλτενμπούργο για τα όσα είπε. Μου άρεσαν τα, τα, τα σχόλια. Δεν, μπορώ να δεν, μπορούμε να, δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω το χρόνο, αλλά αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτήν την έκθεση είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν επιπλέον κίνδυνοι. σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Οπότε δηλαδή θα ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας πριν να προβούμε σε υποσχέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειες απλοποίησης. Είναι το πρώτο κεφάλαιο που μπορούμε να επιτύχουμε συμβιβαστική. Τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν αναφερθεί και ότι αυτά είναι αντιφατικά με την πολιτική συνοχή. Εγώ δεν νομίζω. Όμως όταν τα χρηματοδοτικά μέσα παρουσιάζονται ως πανάκια για τις περιφέρειες, εγώ δεν νομίζω πως ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δούμε και τη γεωγραφική κατανομή των μέσων αυτών, γιατί κατά τη γνώμη υπάρχει ε, έλλειψη ισορροπίας και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Βεβαίως, η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη είναι ένας μηχανισμός που ωφελεί πολλά κράτη-μέλη, αλλά όλα τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, δεν χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής. Αυτά έχω να πω για σήμερα. Ευχαριστώ, και, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ε, και ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Αυτή είναι η συζήτησή μας. Λοιπόν, με βάση την έκθεση που υποβλήθηκε, ξέρουμε πως υπάρχει πρόβλημα με το για την υποβολή των τροπολογιών. Εγώ θα σας προτείνω μια ημερομηνία που μας επιτρέπει να ψηφίσουμε για την έκθεσή μας το Δεκέμβριο. Πράγμα που είναι και το αρχικό πλάνο μας ως Επιτροπή, έτσι δεν είναι, μάλιστα. Λοιπόν, έχοντας υπόψη ότι μπορούμε να ψηφίσουμε στις 3 Δεκεμβρίου, το αργότερο που μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες είναι 22 Οκτωβρίου. να διατηρήσουμε την ημερομηνία της ψηφοφορίας και έτσι δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε κάποιες από τις ομάδες για τις τροπολογίες. «22 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, λοιπόν, προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ε, θα σταματήσουμε τη συνεδρίαση. Ναι, κυρία Κρέλ, ναι, μια σύντομη παρατήρηση. Ξέρω και περιμένω πολλές τροπολογίες, αλλά παρακαλώ, συνάδελφοι, όλοι μας είμαστε βουλευτές και γνωρίζουμε ότι έχουμε σύντομα προεκλογική εκστρατεία, όμως παρακαλώ, δεν είναι ανάγκη κάθε συνάδελφος να να υποβάλει χωριστά και μονομένα τροπολογίε. Αν συνομιλήσετε με τους συναδέλφου του σας, ίσως θα μπορούσατε από κοινού να υποβάλλετε τροπολογίε. Αυτό είναι μία μου παρατήρηση, παράκληση και το δεύτερο είναι Θέλω να σας ζητήσω να μην καταθέσετε όλες τις τροπολογίες που θα εισάγουν αργότερα τα κράτη-μέλη στους τριμερείς, γιατί αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική μας θέση πολύ. Παρακαλώ σκεφτείτε το αυτό και να είστε λίγο πιο αισιόδοξοι ότι έχουμε ισχύ ως βουλευτές. Ναι, ευχαριστώ. Είμαστε πολύ ισχυροί βουλευτέ. ναι. Ε, ε, κύριε Νόβακοφ, και εσείς σε δύο λεφτά. Ναι, έχετε δίκιο ότι υπήρχε το θέμα της προθεσμίας. Αυτό δεν έχει να κάνει με κανένα περιορισμό προς τα ε, συναδέλφους. Απλά να τους θυμίσω ότι τελευταία φορά το CPR πήρε δύο χρόνια. Τώρα είχαμε τρεις μήνες με τον Αύγουστο μέσα. Είμαστε σε μια καλή θετική συγκυρία, οπότε να μην το χάσουμε, να μην τις παταλήσουμε με μαχρονοβόρες διαδικασίες. Πιστεύω ότι θα βρούμε κοινό έδαφος στις συμβιβιστικές, ό,τι τροπολογίες και συμβουβάλλεται. Παρακαλώ λοιπόν να ε, δουλέψουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Αγαπητοί συνεισηγητές, να είστε βέβαιοι, δεν θα σας αφήσουμε μόνο σας. Θα σας υποβάλουμε τροπολογίες και θα σας στηρίξουμε στην αναζήτηση συμβιβαστικών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που κάνατε μέχρι τώρα. Τώρα όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτή τη συζήτηση. 22 Οκτωβρίου προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Κλείνει η σημερινή μας συνεδρίαση και αύριο το πρωί έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Κοτέρ. Με χαρά θα σας δω και πάλι όλους εκεί.